Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, σα προτείνω να αρχίσουμε τι εργασίε σα. Έχουμε μερικά ραβοκαθέσει. Περιέργω δεν έχουν έρθει όλοι. Αυτό τι σημαίνει. Ότι η μέρα του θερινού ηλιοστασίου γιορτάζεται ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες. Πάντως, σας προτείνω καταρχήν την έγκριση μιας διάταξης. Αν δεν διαφωνεί κανένα, θεωρώ ότι είναι κρίθη. Όσον αφορά τι ανακοινώσει του Προέδρου, έχετε στο κόμπο News τις πληροφορίες για τις διαθέσιμες γλώσσες. Η συνεδρίασή μας, όπως και όλες μας συνεδριάσεις, περνάνε στο web streaming, στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τη συνέχεια που δίνεται στην κοινή αντιπροσωπεία που στείλαμε στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης από κοινού, σε επίπεδο κοινοβουλίου την περσμένη εβδομάδα εγκρίναμε ένα ψήφισμα για την κατάσταση στα παρισνιακά εδάφη, ιδίω στη Γάζα. Ιδίω με αυτό που έγινε αμέσω τα που πήγαμε εκεί. Στι 5 Ιουλίου, 7 με 8.30 το βράδυ, θα σα πούμε σε πιάτσα οι τρει αυτέ επιτροπέ που τους αφορά το ίδιο πρόβλημα θα έχουν μια κοινή συνεδρίαση στην οποία θα γράψουν ο κύριο Τζον Γκέινγκ που είναι ο, ο διευθυντής του UNNWRA ε, ε, του οργανισμού αυτού του ΟΗΕ που έχει το γενικό του επιτελείο στην ε, Γάζα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ικανός και μπορέσει να παρουσιάσει την κατάσταση επί τόπου. Γνωρίζω ότι η UNRWA είναι ένας από τους οργανισμούς που διαχειρίζεται ένα τμήμα των πιστώσεων που ε, προβλέπει ο προβλησμός της Ένωσης για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. 13 και 14 Ιουλίου, ιδίω μάλλον στι 13 το απόγευμα, θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Προπολογισμών με τον Πρωθυπουργό τη Παλαιστινιακή Αρχή, τον κ. Σαλαμφαγιάτ. Πρόκειται για μια προσωπικότητα που συναντήσαμε επί τόπου και θα μπορέσουμε μαζί του να δούμε πού βρίσκονται η κατάσταση και ποιες είναι οι ανάγκες των, της Παλαιστινιακής Αρχής όσον αφορά την πολιτική κατάσταση και τους όρους κατά τους διαχειρίζονται τους πόρους. Κατόπιν. Όσον αφορά το σημείο 4, το ανακοινώσεων του Πρόεδρου, η πολιτική συνοχής, ο ειδικός ε, ε εισηγητή, πολυδυναμικό τη τη που απουσιάζει αυτή τη στιγμή, έχει προετοιμάσει κάποιου πίνακε με τα τελευταία στοιχεία εφαρμογή τη πολιτική συνοχή. Οι πίνακε αυτοί υπάρχουν στο φάκελο υπό τον αριθμό 22. Όσον αφορά την εφαρμογή του προπολογισμού 2010, θα ήθελα να σας πω ότι λάβαμε τα τελευταία στοιχεία ημερομηνίες 8 Ιουνίου. Τα στοιχεία αυτά είναι η μας στο διαδίκτυο του Κοινοβουλίου, στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, εκεί που αναφέρεται ο Κόμπο News. Και τέλος πήραμε ένα νέο διορθωτικό προπολογισμό 2010 όσον αφορά τις ανάγκες πιστώσεων για τη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερική δράσης. Πρόκειται τον 6 ερθωτικό προπολογισμό ε, του 2010 και θα πρέπει σε λίγο στους συντονιστές να συμφωνήσουμε όσον αφορά το ποιος θα αναλάβει την έκθεση για το θέμα αυτό. Αυτό σχετικά με τι ανακοινώσει του Προέδρου. Σημείο 3 τη σημερινή διάταξη. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 27η και 28η Απριλίου. Σα έχουν δυναμηθεί τα πρακτικά αυτά. Εάν δεν υπάρχει διαμαρτυρία με θα θεωρήσουμε ότι ενεκρίθησαν. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 4. Όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού 2011 και την θέση του Κοινοβουλίου πάνω σε αυτό. Η συγγετριά μα Σιδόνια έχει ένα έγγραφο εργασία που θα μα το παρουσιάσει. Παρακαλώ, Σιδόνια, έχετε το λόγο. Ε, e, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. αυτό το έγγραφο εργασίας το προετοίμασα στα πλαίσια του προϋπολογισμού 2011. Στόχος αυτού του εγγράφου εργασίας είναι να αναλύσω σε βάθος το πώς λειτουργούν τα προγράμματα για την νεότητα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Έχετε όλοι νομίζω συνειδητοποιήσει ότι τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεότητα και την παιδεία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και για μένα φυσικά. Και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη την οποία μου δώσατε κατά τη διάρκεια της τελευταίας Ολομέλειας όπου μπορέσαμε να τονίσουμε μία από τις προτεραιότητες την οποία οποία είχαμε καθορίσει για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά για την νεότητα θα γίνουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον Ιούνιο και γι' αυτό σε αυτό το έγγραφο εργασίας προσπαθώ να εξετάσω σε πιο, με πιο λεπτομερή τρόπο το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτασης των νέων. Έχει συνταχθεί το κείμενο εργασίας αυτό στην αγγλική γλώσσα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλές μεταφραστικές δυνατότητες στη διάθεσή μας και σας ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να παραδώσω το έγγραφο αυτό και στις υπόλοιπες γλώσσες. Ελπίζω όμως στα αγγλικά να μπορέσουμε όλοι να εργαστούμε ικανοποιητικά. Να σας παρουσιάσω τις βασικές αρχές. Έχω, θα έλεγα, διαιρέσει το έγγραφο σε δύο τμήματα. Καταρχάς, τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται άμεσα από τον προϋπολογισμό και δεύτερη κατηγορία είναι τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται έμεσα για τα άμεσα χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε τη διαβίου κατάρτιση. Πρόκειται για μια τεράστια θα έλεγα σε μέγεθος γραμμή του προϋπολογισμού. Υπάρχουν εδώ τα γνωστά προγράμματα κομένιους εράσμους, και ό,τι άλλο έχει σχέση με την ανώτερη εκπαίδευση. Έχουμε το Λεωνάρτο Νταβίντσι για επαγγελματική κατάρτιση και γενικότερα άλλα προγράμματα για οριζόντια λεγόμενα για ενηλίκους εκπαίδευση καθηγητών, διδασκόντων αποστολή διδασκόντων στο εξωτερικό, διδασκαλία ξένων γλωσσών, γενικά πολύ φιλόδοξα και διαφοροποιούμενη ε, στο εσωτερικό της γραμμή του προϋπολογισμού που δεν καλύπτει μόνο τους νέους, αλλά και άλλα θέματα τα οποία καλύπτονται από τις τρεις λέξεις νεότητα, εκπαίδευση, κινητικότητα. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το Erasmus Mundus. Υποστηρίζουμε μέσω του Μούντους ε, τα συστήματα εκπαίδευσης σε άλλες χώρες και βοηθάμε, ευνοούμε την κινητικότητα των σπουδαστών. Βέβαια αυτό το πρόγραμμα είναι μικρότερο Το έχουμε χρησιμοποιήσει και για την υποστήριξη μη θεσμικών μορφών εκπαίδευσης. Μορφές εκπαίδευσης που αποκτούν νέα σημασία στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Ξέρετε ότι υπάρχουν και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο κάποια τμήματα που αφορούν την κινητικότητα των ερευνητών. Και εκεί υπάρχουν τμήματα δηλαδή τα οποία μας ενδιαφέρουν. Σχετικά με τα δημοσιονομικά μέσα τώρα στο δεύτερο τμήμα τα οποία χρηματοδοτούν έμεσα. Έχουμε το Progress, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και με μονομένες δράσεις και μικρότερα προγράμματα που ε, χρηματοδοτούν τους νέους σαν παράδειγμα γεωργούς που χρηματοδοτούνται από το δεύτερο τμήμα του προϋπολογισμού. Τα προγράμματα αυτά έχουν γίνει αντικείμενο περιγραφής ε, αναλυτικά στο κείμενο εργασίας και δεν χρειάζεται να σας τα παρουσιάσω αναλυτικότερα. Ε, η απορρόφηση αυτών των προγραμμάτων, των δυνατοτήτων των οικονομικών δηλαδή που παρέχουν φτάνει σχεδόν το 100%. Υπάρχει δηλαδή εμπειρογνωμοσύνη πλέον σχετικά με τα προγράμματα αυτά. Λοιπόν, εκπαίδευση, νεότητα και κινητικότητα. Υπάρχουν και κάποια άλλα μέσα που εξυπηρετούν αυτούς τους τρεις στόχους από το τμήμα 2 και το πέμπτο κεφάλαιο που ασχολείται με θέματα γεωργίας πιο συγκεκριμένα. Φυσικά στο έγγραφό μου περιγράφω και τις διάφορες υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή των δράσεων των σχετικών με την κινητικότητα και την εκπαίδευση. Έχουμε την Υπηρεσία για την Επαγγελματική Κατάρτιση και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Κατάρτιση. Είναι εξωτερικές υπηρεσίες, αποκεντρωμένες λεγόμενες υπηρεσίες, και υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες εξωτερικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Στο κείμενο εργασίας υπογραμμίζεται επίσης το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα η ημερήσια διάταξη σε εισαγωγικά 20-20 άπτεται των νέων ιδιαίτερα. Περιγράφω κάποια επιπλέον προγράμματα όπως το γνωστό Youth and Move και θα υπάρξουν και άλλες ιδέες ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν σύντομα σχετικά με τα κύρια τουλάχιστον προγράμματα που συναποτελούν τον στόχο 2020. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σας έχω ήδη πει τα προγράμματα τα σχετικά με την κινητικότητα, την εκπαίδευση και την νεότητα παράγουν προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Βοηθούν τους ενήλικες αλλά και τους νεότερους να αποκτήσουν θα έλεγα ένα ευρωπαϊκό πνεύμα και με τον τρόπο αυτό τα προγράμματα βοηθούν την ευρωπαϊκή ιδέα εκτός από τους πολίτες. Είναι προγράμματα τα οποία θα χαρακτήριζα και ιδιαίτερα οικονόμα σε σχέση ε, με, ε, με το σύνολο των δαπανών. Αν σκεφτεί κανείς πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που καλύπτονται από τους στόχους αυτούς, θα δει ότι τα ποσά και δεν είναι μεγάλα και δαπανώνται αποτελεσματικά και γενικά είμαι στη διάθεσή σας πάντως αν θέλετε για περισσότερες πληροφορίες. Σε ευχαριστώ Συντόνια για ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο. Είναι για πρώτη φορά που αποπειραθήκαμε να συγκεντρώσουμε στο συγκεκριμένο κείμενο το σύνολο των προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες της νεότητας ε, με την ε, ευρία έννοια. Όπως είπε η συγγήτρια, είμαστε πάντα στα πλαίσια της γραμμής 2020 όπως υιοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στα πλαίσια του ψηφίσματος που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 2020. για το ποσοστό δραστηριότητας και του συνόλου του πληθυσμού και των νέων έχουμε θέσει νέους στόχους έτσι ώστε το 40% των νέων να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο κατάρτισης που να καλύπτεται από την ανώτατη εκπαίδευση και να έχουν διπλώματα ανώτατης εκπαίδευσης και έχουμε και αρκετούς άλλους φιλόδοξους στόχους στα πλαίσια του 2020, της στρατηγικής 2020. Ε, να προσθέσω εδώ μια προσωπική πληροφορία. Στο Μπορντό, στην εκλογική μου περιφέρεια, την Παρασκευή, φιλοξενήσαμε μια συνάντηση των ε, Γάλλων και Γερμανών βιοτεχνών. Κάθε τρία χρόνια τα βιοτεχνικά επιμελητήρια που εκπροσωπούν αυτούς τους εργαζομένους της Γερμανίας και της Γαλλίας συναντώνται, ανταλλάσσουν πληροφορίες και επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές από κοινού. 11 χώρες, σε 11 χώρες μάλλον, οι βιοτέχνες έχουν ένα καθεστώς που αναγνωρίζεται από τον νόμο και έχουν επαγγελματικές οργανώσεις που διαχειρίζονται τα επαγγέλματά τους και ισχύει αυτό και για τη Γαλλία και τη Γερμανία. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ένα πρόγραμμα όπως το πρόγραμμα Λεωνάρντο που είναι θα έλεγα για τους νέους εργαζομένους του Εράσμους για τους φοιτητές. Είδαμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα Λεωνάρντο δεν δούλευε καλά και είχε πολύ χαμηλότερα ποσοστιαία αποτελέσματα από το Εράσμος. Στην γαλλογερμανική περίπτωση καταλήξαμε σε μια διαφορετική επιλογή ανταλλαγής 20 με 30 χιλιάδων βιοτεχνών Γάλλων και Γερμανών που μετακινούνται στα πλαίσια ενός διμερούς μηχανισμού που ισχύει εδώ και 40 χρόνια της, Αγγλο... της γαλλογερμανικής υπηρεσίας νεότητας. Σας το λέω αυτό ε, όχι για να δείξω ότι υπάρχουν ειδικέ ανάγκες ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά γιατί τελικά βρήξαμε, βρήκαμε ένα σύστημα που επιτρέπει τις ανταλλαγές των επαγγελματιών ανάμεσα στις δύο χώρες αυτές. Τα αποτελέσματα αυτών των ενταλλαγών μου δίνουν να καταλάβω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το οποίο κάνει το Λεωνάρντο στο σύνολο των 27 χωρών κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντα 2020 και για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες μας προτείνει η συγγήτρια με την υποστήριξη του συνόλου του Κοινοβουλίου που υιοθέτησε το, την εντολή διαπραγμάτευση την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Συντονία για το τόσο σημαντικό αυτό έγγραφο. Είναι πολύ χρήσιμο. που έχουμε σε ένα κείμενο όλες τις πληροφορίες που είναι κανονικά διασπαρμένες σε διάφορες γενικές διευθύνσεις και υπηρεσίε. Έχω ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Το σχόλιο είναι ότι υπάρχει ένας τομέα που θα πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε, δηλαδή η μετάβαση από τα εκπαιδευτικά συστήματα στην αγορά εργασία. Δεν υπάρχει πολλά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λαμβάνουν υπόψη αυτό το σημείο. Το κοινωνικό ταμείο κάτι κάνει, αλλά μόνο για τι λιγότερο ευνοημένε περιοχέ. έχουμε ε, μία πάση πιλότου το έρασμος για τους νέους επιχειρηματίες και θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα για να γίνει ένα μόνιμο πρόγραμμα στο μέλλον. Αλλά δεν αναφέρεται νομίζω αυτό στην έκθεση. Δεύτερη ερώτηση. Ορισμένα αυτά τα προγράμματα αυτά είναι εστιασμένα και στην νεολαία αλλά και στο ευρύτερο κοινό όπως το κοινωνικό ταμείο ή άλλα προγράμματα στα οποία έχουν πρόσβαση άνθρωποι που είναι πάνω από 35, κάτω από 35 κλπ. Μπορούμε να υποδιαιρέσουμε αυτά τα κονδύλια γιατί αλλιώς δίνουμε την εντύπωση ότι θα περνούν περισσότερα χρήματα από εκείνο που πραγματικά είναι διαθέσιμα για την νεολαία. Το ίδιο και για την Μαρή ε, Curie. Υπάρχουν διάφορες υποτροφίες. Υπάρχουν μετά δύο υποτροφίες για άτομα που είναι πιο νέα. Θα μπορούμε λοιπόν ίσως να διακρίνουμε ποιες είναι οι πραγματικές, ε, τα πραγματικά κονδύλια σε αυτά τα προγράμματα που ε, έχουν σαν στόχο την ολία και ποια όχι. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. έχει ο Σαλβαντόρ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έγγραφο αυτό, το οποίο καταρχήν είναι πάρα πολύ χρήσιμο πέραν ε, της ε, ακαδημαϊκής της ε, αξίας, της ερευνητική δουλειάς που έκανε, ούτως ώστε να μπορέσουμε εδώ να αποτυπώσουμε όλα όσα κατά κάποιο τρόπο έχουν να κάνουν με την κάθε πολιτική που αφορά τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως αυτό αφορά κάποια αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού τα οποία θα πρέπει να τα τροποποιήσουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε τα υπεσχημένα, να τηρήσουμε αυτήν την διαπραγματευτική εντολή για την συντόνια της 30ης Ιουνίου. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με την ε, μεταβολή των κονδυλίων για τον Σεπτέμβριο. Επίσης θέλω να τονίσω αυτή την σχέση την οποία τονίζει και η συγκήτρια όσον αφορά Σαλβαντόρ, Σαλβαντόρ λέει ο πρόεδρος, μου λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν περνάει η μετάφραση, η διερμηνία. Να προσπαθήσω. Α, τώρα, τώρα, τώρα δουλεύει. Στα, στα Ουγγρικά ακούτε? Μετάφραση προς τα Ουγγρικά λειτουργεί. Ο βουλευτής μιλά εκτός μικροφώνου και δεν ακούει, δεν το έχει ανάψει, δεν ακούγεται. Βεβαίω και είναι κατανοητό, σε οποιαδήποτε γλώσσα, έτσι και λέει ο Σαλβαντόρ, λέει ο πρόεδρο. Για που ξαναπροσπάθησε Σαλβαντόρ. Να συνεχίσω στα αγγλικά κατευθείαν ή στα ισπανικά. Καλά, τέλο πάντων. Θα συνεχίσω στα ισπανικά που τα καταλαβαίνετε ίσως και καλύτερα και επομένω ήθελα να σας πω ότι μου ήλκησε την προσοχή η σχέση αυτή που αναδεικνύει η συγγήτρια μεταξύ αυτών των flagship της ναυαρχίδας της πολιτική του 2020 και των πολιτικών για την νεότητα οπότε κανείς θα έλεγε ότι ε, η βασική τέτοια ναυαρχίδα του ΣΥΠΗΝ είναι αυτό που περιγράφεται σε αυτή την πρωτοβουλία cuatro, eh, dos, tres, otras tres eh, eh flagships eh, donde... Eh, έχουμε και τις άλλες ναυαρχίδες, τα άλλα θέματα τα βασικά όσον αφορά τα προγράμματα για την νεολαία και την νεότητα που θα πρέπει και αυτό να καλυφθούν και όταν έρθει η ώρα η συντόνια να κάτσει και να λάβει υπόψη αυτό το οποίο είπαμε για να δούμε πώς και οι άλλες πρωτοβουλίες ε, μπορούν να οδηγήσουν σε μια καινούργια ατζέντα ψηφιακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα έχουμε και καινο, πολιτικές καινοτομίες, πώς όλα αυτά θα περάσουν μέσα από τα, τα, τα, προγράμματα της πολιτικής για την νεότητα και τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι μια σαφής πρεκοδότηση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σαλβαντόρ και δίνει το λόγο κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, όπως και η Συντόνια, θεωρώ ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα όσον αφορά τις πολιτικές νεότητας και έρευνας και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, έχουμε αυτή την προβληματική ε, πολιτική του 2020, οπότε και έχουμε την ισόβια κατάρτιση, ε, θέματα που αφορούν το κοινοβούλιο, κινητικότητα των νέων, έρευνα, που θα πρέπει όλα αυτά να είναι οι πυλώνες για την στρατηγική για το 2020. Εγώ θα ήθελα επίσης αυτή την προσέγγιση να την επικροτήσω και εάν δείτε την απασχολησιμότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη θα διαπιστώσετε ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα του πώς θα έχουμε περισσότερους πεπαιδευμένους και κατηρτισμένους, μια που τώρα έχει αλλάξει η αγορά ε, έχουμε εξελίξει και τη τεχνολογική αλλά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο στον τομέα της παιδείας και από νωρί να μπορεί κανείς να έχει τις δεξιότητε που πρέπει, οπότε να συνειδητοποιηθεί ότι η ισόβια κατάρτιση είναι κομμάτι της ζωή μα. και ότι τελικά δεν αφορά μόνο τους νέους αλλά ότι είναι κομμάτι της διαδρομής της ζωής μας αυτά, τα οποία θα πρέπει να τα κάνει στη ζωή του αυτή τη, την, της, της περίοδου της κατάρτισης. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς απαιτείται, ποιες είναι οι νέες προκλήσεις και να επενδύσουμε επομένως περισσότερα στην παιδεία και αυτό θα μας αμύψει από πλευράς ανταγωνιστικότητας. Επίσης, να προχωρήσουμε σε κάποια συνεννόηση με τα εθνικά κοινοβούλια. Πρόεδρε, κύριε Λαμασούρ και εσείς συμφωνείτε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο τόσο ώστε να βγούμε κερδισμένοι συνεννόηση εν ώψη για το 2020, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και σε επίπεδο Συμβουλίου και να το συνεννοηθούμε με τα εθνικά κοινοβούλια γιατί είναι προς το συμφέρον όλων. Θα πρέπει 3% του εθνικού προπολογισμού να πάνε στην έρευνα και στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχουμε πετύχει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αλλά δεν είναι καθόλου σαφές εάν θα πετύχουμε περισσότερα με την συνθήκη, τη στρατηγική της Λισαβόνας, άρα να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε και στις λεπτομέρειες του το πώς θα περάσουν αυτά τα θέματα που είναι πανεπιστημιακού ενδιαφέροντος και συμφέροντος μέσα από το διάλογο με Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Φέρουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συμφωνώ 100% με όσου ήδη έλαβαν το λόγο, πολύ αξιόλογο αυτό το έγγραφο. Είναι καλύτερη αποτύπωση του, τοπίου που έχουμε μπροστά μας, που έχω δει ποτέ. Και αποδεικνύει αυτό το οποίο είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες για το ψήφισμα για το ότι το, το, το, θέμα των νέων δεν είναι μόνο γεννητικότητα. Έχουμε και κοινωνικά θέματα και πολιτιστικά που είναι εξίσου σημαντικά. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό το έγγραφο αποδεικνύει αυτό το οποίο λέγαμε. Πρόκειται για ένα θέμα όπου ίσως δεν έχουμε όλα τα δεδομένα τα οποία χρειαζόμαστε, δηλαδή το κοινωνικό ταμείο και ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν έχουμε σαφές το τι χρειάζεται γι' αυτό και χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες που θα πρέπει να μας τις δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι για την τελευταία παράγραφο να σας πω, εκεί που αναφέρει η συγγήτρια ότι θα πρέπει να έχουμε πρικοδότηση για τέτοιου είδους μέτρα εν ώψη τη συζήτηση του Οκτωβρίου για τον προπολογισμό θα κατεβάσει συγκεκριμένε προτάσει η συγγήτρια για το πώ θα πρέπει να ενισχύσουμε τα αντίστοιχα κονδύλια για να πετύχουμε του στόχου που θέλουμε. Όμω δεν υπάρχει και μεγάλο περιθώριο βελτιώσεων. Άρα, ιδίω όσον αφορά το 1α και το 3β, από ό,τι βλέπω, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Η συγγήτρια εδώ ξεκίνησε κάποια ανάλυση. Έχουμε αυτό το 5% της ευελιξίας. Ήδη έχουμε κάποια κονδύλια σε αυτούς τους τίτλους τα έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά επί τη βάση των δημοσιονομικών προοπτικών και έχουμε δεσμεύσεις κατά προτεραιότητα και σε άλλα θέματα από Επιτροπή Απασχόλησης, από Επιτροπή Πολιτισμού και για προπαρασκευαστικές πράξεις και για προγράμματα. Άρα πώς όλα αυτά θα συντονιστούν η συντόνια. Νομίζω ότι άρχισε εδώ πέρα να σκέφτεται περικοπές. Γιατί χωρίς περικοπές δεν μπορώ να διαπιστώσω πού θα βρούμε το περιθώριο να βελτιώσουμε τα κονδύλια αυτά. Τι λέτε. Σε ευχαριστώ, Γκόρεν. Ίγκα. Ευχαριστώ. Ο πένεσαν τη Συντονία μπορώ και εγώ να το κάνω. Αλλά αυτό που μου λείπει είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας γιατί εμένα με έκανε να απορρίψω πόσα προγράμματα άπτονται του θέματος της Νοηλέας και θα ενδιαφέρον να δούμε πόση διαχείριση χρειάζονται αυτά τα διάφορα προγράμματα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του εγγράφου της Ιδονίας θα μπορούσε να μας ε, ε, δώσει κάποια στοιχεία για το πόση διαχείριση χρειάζονται τα προγράμματα αυτά. Στην αρχή της ε, νομοθετικής ε, περίοδου είχα ρωτήσει κάτι παρόμοιο για το θέμα της ε, διαχειριστικής προσπάθειας. Βέβαια τα στοιχεία που έχουμε εδώ είναι πολύ ψηλά. Θα ήταν καλό να είχαμε κάποιες συγκεκριμένε πληροφορίες. Γι' αυτό θέλω παρακαλώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο πρόεδρος, η Ίγκε έθεσε το δάχτυλο από τον τύπο των ήλων σε κάτι που δεν είναι το πραγματικό πρόγραμμα, ότι σε αυτού του τύπου τα οριζόντια προγράμματα εμπλέκονται περισσότερες στις μία γενικές διευθύνσεις κομισιών και περισσότεροι επίτροποι του ενός. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος αντιφάσεων, επικαλύψεων, προβλημάτων. Δεν ξέρω, κατά πόσο ο Γενικό Διευθυντή ε, που μα θυμά με την, παρουσία με την παρουσία του θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Αλλά προηγουμένω θα δώσουμε το λόγο στον Τζέιμ Έλλε. Παρακαλώ, Τζέιμ. Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο αυτό και σε μια γενική προσέγγιση. Αυτά τα έγγραφα που έχουμε για την Ευρώπη το 2020 για την νεολαία, κινητικότητα της νεολαίας. Όλα αυτά σχετίζονται με το πώς πετυχαίνουμε με τις νέες τεχνολογίες τις απαραίτητες ικανότητες. Ε, μέχρι το 2015 95% των θέσεων απασχόληση λένε χρειάζεται, θα, έχουν ένα παράγοντα ε, αλλά μόνο το 30% σήμερα είναι ενήμεροι. Θα υπάρχουν λοιπόν προβλήματα. Τόσο περνάει τα προγράμματα αυτά και τονίζουμε τι νέε τεχνολογίε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε εκ των υστέρων τι έχουμε πετύχει και βέβαια και πού θα πεσαίνουν τα χρήματά μα. γιατί εγώ βλέπω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχίσει και για το 2011. Δεν θα μπορούμε να ξεχάσουμε ότι τα κράτη-μέλη περικόπτουν τους προπολογισμούς τους. Η Ιταλία, η Γερμανία, η δική μου χώρα, όλοι περικόπτουν τους προπολογισμούς τους. Ε, νομίζω αναφέρατε τις δυσκολίες που θα υπάρξουν προσεχώς, κύριε Πρόεδρε, εσείς την περασμένη φορά που μιλήσατε στην Επιτροπή Πολιτισμών. Ίσως πολλοί συνάδελφοι να μην συμφωνούν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά μέχρι τα τέλη τη διαδικασίας αυτό θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί οι πιέσει ε, στα κράτη-μέλη αυτό θα μα πείσουν ότι χρειάζεται. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε το προπολογισμό 2011 όταν περιμένουμε ότι θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα για το προπολογισμό το 2012, 2013, 2014. Πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο πού βρισκόμαστε στη στιγμή και η δυνατότητα δημιουργίας πλειοψηφιών είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Merci, merci James. Ευχαριστώ James. Πράγματι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα των δημοσιονομικών επιλογών και των πιστώσεων που θα πρέπει να ψηφιστούν για το 2011 λόγω των τελευταίων εξελίξεων. Έχω εμπιστοσύνη στην αντιπροσωπεία του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του τριμέρους διαλόγου για να μας προσγειώσει. Ας ελπίσουμε ότι η προσγείωση δεν θα είναι ιδιαίτερα βίαιη το θέμα είναι ανεξαρτήτως του ύψους των ποσών να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Μπορούμε να κάνουμε μειώσεις σε όλα αν θέλετε. Από την άλλη μπορούμε να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε κάποια προγράμματα τα οποία μας φαίνονται πιο σημαντικά. Η κάθε κυβέρνηση αυτά κάνει. Πρόκειται για μια προσπάθεια χρήσιμη για όλους. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής θα μεταφέρει τις απόψεις της διεύθυνσής του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ συνοπτικός. Τρία σημεία. Πρώτον, να συγχαρεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εισηγήτρια σχετικά με την ποιότητα της εκθέσεως που υπευλήθη. Έχει γίνει πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και θα ωφελήσει πολύ στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να προκαλέσω και την προσοχή των μελών για δύο έγγραφα που ήδη έχουν διανεμηθεί. Το πρώτο διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Monitoring Group 4 Μαΐου και απαντά θα έλεγα σε πολλές ερωτήσεις, ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τα επιμέρους προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες των νέων, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες των νέων. Ένα δεύτερο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτό το οποίο έχει ημερομηνία 7 Ιουνίου και αφορά τα θέματα στα οποία δεν δόθηκαν απαντήσεις στο παρελθόν περιλαμβάνει νομίζω αρκετά συγκεκριμένες υποδείξεις για τα προγράμματα που καλύπτουν την νεότητα και για τις δυνατότητες που παρέχει στον συγκεκριμένο τομέα το κοινωνικό ταμείο. Τρίτη παρατήρηση, απαντώντας εδώ και στο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε για το διοικητικό κόστος. Δεν πρόκειται για μια βέβαια ευθυνή θα έλεγα απόπειρα και αποστολή. Το διοικητικό κόστος εξαρτάται, καταλαβαίνετε, από το μέγεθος της ε, πολιτικής παρέμβασης και της πολιτικής που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε είναι σαφές ότι θα έχουμε σύντομα ένα επίπεδο λεπτομέρειας το οποίο σε αυτή τη φάση δεν είναι αντίστοιχο με την επιθυμία της κυρίας Γκρέσλε. Ευχαριστώ, η συγκήτρια έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που πήρατε το λόγο Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που είπατε ότι είναι καλό το κείμενο, γιατί εγώ είχα πολλά προβλήματα με το κείμενο αυτό, δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, γιατί τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχουμε ένα καλό έγγραφο δεν τα είχα στη διάθεσή μου. Θα σας πω δηλαδή και ποιες είναι οι αδυναμίες της διαδικασίας αυτής. Το θέμα είναι λοιπόν ότι για να έχει κανείς ε, καλά δεδομένα για το σύνολο των συμμετεχόντων, την ηλικία των συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα, τους καρπούς δηλαδή της προσπάθειας, το κατά πόσον έχουν υπάρξει βελτιώσεις στις εκπαιδευτικές τους δυνατότητες ή να έχουμε μια εκτίμηση κατά κεφαλήν σε εισαγωγικά κόστους. Δεν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα έχει, οι εθνικές υπηρεσίες δεν τα έχουν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ θέλει ολόκληρο ερευνητικό πρόγραμμα για να τα έχει όλα αυτά. Δεν έχουμε συνεπώς τα μέσα τα οποία θα μας επέτρεπαν να δώσουμε αξιόπιστες πληροφορίες για τα προφίλ, τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, την ηλικία τους, την εκπαιδευτική τους κατάσταση. Έχουμε μόνον επιμέρους διάσπαρτα στοιχεία αυτής της προσπάθειας. Γνωρίζουμε πράγματι πάρα πολύ λίγα για το τι μπορούμε να κερδίσουμε από το πρόγραμμα αυτό. Ίσως αν μου επιτρέψετε να περάσω σε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που προσπάθησα να πετύχω σαν εισηγήτρια και το έχω ήδη πει στην συνάντηση που είχαμε τον μήνα Μάρτιο αποφάσισα θα έλεγα να ακολουθήσω τρεις προτεραιότητες. Νεότητα, εκπαίδευση, κινητικότητα. Έτσι ώστε να μπορέσω να ξεπεράσω το πρόβλημα του ποια είναι τα προγράμματα που ωφελούν τους νέους. Είναι δύσκολο πολλές φορές να είναι κανείς βέβαιος και ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί, αν συμμετέχοντες ή ωφελούμενοι από ένα πρόγραμμα είναι 26 ετών, 30 ετών, 36 ετών ή λιγότερο. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη σημασία δεν έχει η ηλικία. Σημασία έχει τα προγράμματα αυτά να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών τη στιγμή από την οποία περνάνε από το εκπαιδευτικό στάδιο στο επαγγελματικό στάδιο. Αυτό έχει σημασία και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται ε, το κριτήριο για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών και όχι το αν θα καλύπτουν ανθρώπους ηλικίας 25, 26 ή κάποιες άλλες. Ένα παράδειγμα της δυσκολίας που αντιμετώπισα. Έθεσα ορισμένες ερωτήσεις στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Επιτροπής. Ποιοι αποφελούνται από το Κοινωνικό Ταμείο Ποιοι είναι αυτοί. Βρίσκουν δουλειά μετά την εκπαίδευση. Πιο εύκολα από αυτούς που έχουν εκπαιδευτεί, έχουν καταρτιστεί. Προσπαθούν να μου δώσουν τις πληροφορίες αυτές, αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι θέμα περίπλοκο, είναι θέμα που αφορά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα εν πάση περιπτώσει και πρέπει να εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο. Το κόστος ε, κατά πολίτη που καλύπτεται από τα προγράμματα αυτά. Πόσο κοστίζει αναπολίτη το πρόγραμμα. Αν το συγκρίνουμε με κάποιον ο οποίος ε, σαν παράδειγμα σε μια νεότερη ηλικία έχει την δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε νέους τομείς. Εγώ έκανα κάποιους υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί μου λένε λίγο πρόχειρα βέβαια ότι τα τοπικά προγράμματα που αφορούν τους νέους, η επαγγελματική κατάρτιση τοπική των νέων είναι φθηνότερη από τις παρεμβάσεις του κοινωνικού ταμείου. Πολύ φθηνότερη. Παρ' όλα αυτά Προσπάθησα να καλύψω όλους αυτούς τους τρεις τομείς τους οποίους προανέφερα, νεότητα, εκπαίδευση και κινητικότητα. Προσπάθησα επίσης να ενσωματώσω και το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Εγώ αν θυμάστε διαμαρτυρήθηκα σε αυτά που είπε ο Λεβαντόφσκι να συμπεριλάβουμε το σύνολο του 7ου προγράμματος πλαισίου στα προγράμματα για την νεότητα γιατί από μόνο του είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένα άλλο πρόβλημα ε, και το οποίο έθεσαν κάποιοι από τους συναδέλφους είναι η καλύτερη και περισσότερη ενημέρωση για τις προτεραιότητες αυτές μέσω μεγάλων προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το Ταμείο Ανάπτυξης στο Περιφερειακό. Αυτές τις πληροφορίες τις περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να μην περιμένετε να έχουμε ξεκάθαρες εικόνες της κατάστασης, γιατί τα δεδομένα που έχουν συλλογεί σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων δεν είναι πλήρη δεν προεβλέπεται να συλλέγονται τα στοιχεία αυτά στο παρελθόν. Θα ζητούνται βέβαια στο μέλλον τέτοια στοιχεία και από τα εξωτερικ, τις εξωτερικές υπηρεσίες. Αλλά είναι λυπή τα στοιχεία και δεν μπορώ να βρω λύσεις στα προβλήματα αυτά σε αυτή τη φάση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η στρατηγική 2020 Πολύ πρόσφατα πριν ξεκινήσω να εργάζομαι γύρω από την συγκεκριμένη αυτή έκθεση πήρα στοιχεία από την Επιτροπή Πολιτισμού, την πρόεδρό της, που με ενημέρωσε αρκετά για τις συζητήσεις που είχαν κάνει και φαίνεται ότι υπάρχουν δύο παράλληλες διαδικασίες. Από τη μία είναι τα υπάρχοντα προγράμματα και από, τη λεγόμενη, και από την άλλη είναι τα λεγόμενα flagships, οι ναυαρχίδες των προγραμμάτων. Προφανώς και χρειάζεται περαιτέρω χρηματοδότηση για κάποια από τα προγράμματα αυτά. Δεν υπάρχει όμως απάντηση στις ανησυχίες αυτές σε αυτή τη φάση. Και εγώ είπα ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην θίξουμε τα υπάρχοντα προγράμματα και να μην βρούμε νέα προγράμματα κατάρτισης γιατί αυτό θα μας αποπροσανατολίσει σε αυτή τη φάση. Για το πού θα βρούμε τις πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων. Είναι ένα θέμα που σας απασχολεί ιδιαίτερα. Συμφωνώ 100% με τον πρόεδρό μας λέγοντας ότι αυτή τη βρώμικη δουλειά κόβοντας δηλαδή ποσά θα τα κάνει το Συμβούλιο. Δεν θα είμαι εγώ ο οποίος θα ξεκινήσω λέγοντας εμείς να κάνουμε μειώσεις. Όχι γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά το συμβόλαιο είναι σαφές ότι θα το κάνει καλύτερα και θα έχουμε τα στοιχεία που απαιτούνται αρκετά γρήγορα στη διαδικασία αυτή από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Θα ήθελα να ενισχύσω τις γραμμές οι οποίες έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι χρήσιμες. Σίγουρα το πρόγραμμα Έρασμος, το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση, Youth in Action, και περιμένω να έχω και feedback από τις εξειδικευμένες επιτροπές ε, να δω πώς ακριβώς ε, οι αρμόδιες αυτές επιτροπές βλέπουν τα πράγματα. Τώρα τα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχω συμπεριλάβει ένα μικρό πίνακα στο παράρτημα υπαρίθμ 1 να τονίσω απαντώντας την κυρία Καρβάλιο ότι η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης μαζί με την Επιτροπή την Κοινοβουλευτική Απασχόλησης εργάζονται για κάτι το οποίο υποστηρίζουμε όλοι νομίζω δεν είναι μυστικό. Είναι το θέμα της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Ε, προετοιμάζεται μία προπαρασκευαστική δράση η οποία σας συνδέεται με το ε, δίκτυο EURES που είναι το δίκτυο συνεργασίας των Εθνικών Υπηρεσιών Απασχόλησης θα, παρομοιάζει, θα προσωμιάζει με το Εράσμους όχι για φοιτητές αλλά για αυτούς οι οποίοι αναζητούν την πρώτη τους απασχόληση. Να μπορούν δηλαδή να πηγαίνουν σε άλλη χώρα της Ένωσης και να ξεκινούν την επαγγελματική τους ζωή. Στην ουσία είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με το έρασμος, αλλά παίρνει μορφή προπαρασκευιστικής δράσης για αυτούς οι οποίοι εισάγονται στην αγορά απασχόλησης. Θα δούμε τι θα απαιτηθεί, θα δούμε τι επιτυχία θα έχει αυτό το πρόγραμμα και τι αποτελέσματα γενικά θα έχουμε. Αυτά. Ευχαριστώ Συντονία σημειώνουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στα πλαίσια μιας πολιτικής που σα στόχο να βοηθήσει την ωραία να βγει η θέση απασχόληση και να ωφεληθεί από τον ευρωπαϊκό χώρο πλήρω. υπάρχουν και τα ένομα μέσα κοινωτική νομοθεσία που διευκολύνει την κινητικότητα φορέντου. Και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω το 2005 υιοθετήσαμε μια οδηγία για την αμοιβαία αναγνώριση των ε, διπλωμάτων ή της επαγγελματική ε, εμπειρίας των ε, τεχνητών. 2005 λέω και πέντε κράτη-μέλη ακόμα δεν την έχουν μεταφέρει στο ιστορικό του κρατικό δίκαιο. Η Ελλάδα το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Γαλλία. Ντροπή είναι. Είναι ντροπή πραγματικά. Να, ας πούμε, μια απόφαση που μπορούμε να πάρουμε λίγο και δεν κοστίζει τίποτα. Αυτό το διαβατήριο επίσης που λέγεται Europass που αποδεικνύει την επαγγελματική εμπειρία που μπορεί κανείς να έχει συλλέξει όταν εργάστηκε σε διάφορε χώρε. Αυτό δεν αφορά μόνο του νέου, αλλά και όποιου εργαζόμενου έχουν εργαστεί σε διάφορα κράτη-μέλη και χρειάζεται κάποια αρχή που έχει το, το κάνει να μπορούν να αποδείξουν ότι εργάστηκαν σε μια χώρα ορισμένο αριθμό χωρών. Και εδώ είναι το αντίθετο. Έξι χώρε περίπου έχουν έχουν ε, υιοθετήσει το Europass και οι άλλες 20 όχι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για δράση υπέρ των νέων, αυτό περνάει από δημοσιονομικέ τάξει, προγράμματα ειδικά που υιοθετούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν επιτάπητο ήδη ηλυμένε αποφάσει, οι οποίε δεν έχουν ακόμα αποκτήσει την ε, πραγματική του σημασία. Σα ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε τώρα το σημείο 4 της σημερινή διάταξη. Έχουμε προβλέψει να περάσουμε τώρα στο σημείο 9 και 10. Πριν περάσουμε στα, στοιχεία, στα σημεία για το προπολισμό 2010. Το σημείο 9 είναι η χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Τομείου Προσαρμογή στην Ο συνάδελφο Μικέλ Πορτά είναι ο εισηγητή. Και έχουμε καλέσει επίσης συνάδελφο της ε, Επιτροπής Απασχολής που είναι αρμόδιος για την γνωμοδότηση από αυτού. Θα έρθει εδώ. Αλλά καταρχήν να ακούσουμε τον εισηγητή μας. Ο κύριος Πόρτας έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω πρόβλημα συζητής μια έκθεση για τη χρηματοδότηση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Τομείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Καταρχήν, όταν ξεκίνησα, δεν είχα καμία προκατηλημένη άποψη. Εγώ είπα ότι θα πρέπει να υπάρχει το ταμείο αυτό και να συνεχίσει να λειτουργεί, να το αλλάξουμε. Δεν ήξερα τι θα πρέπει να γίνει. Άρχισα λοιπόν από το μηδέν, όπως σας λέω. η ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται αυτό το ταμείο είναι καλή. Αν εξετάσουμε τα 2,5 χρόνια κατά, κατά τα οποία λειτουργήσε αυτό το Ταμείο από το 2007 στο Μάιο του 2009 δεν πρέπει κανένας να πει ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Οκτώ κράτη-μέλη μοναχά ζήτησαν πόρους από το Ταμείο αυτό. Δεν έχουν εμπλακεί πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Αλλά τους 11 αρχικές προτεραιότητες που υπήρχαν τα χρήματα που επιστράφησαν ήταν έτσι τάξης του 40% από τα χρήματα δηλαδή που καταρχήν καταβλήθησαν επιστράφησαν. Λοιπόν, καλή ήταν η ιδέα, το Ταμείο όμως δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Μετά το Μάρτιο του 2009 υπάρχει ένας νέος κανονισμός που διέπει αυτό το ταμείο. Ένα χρόνο δηλαδή περίπου λειτουργεί υπό τον νέο κανονισμό και αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε γιατί ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου αυτού κανονισμού μπορούμε να πούμε ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ η λειτουργία του Ταμείου και πέτυχε πολύ περισσότερα. Και ένας λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να σταματήσουμε, να, να πάσει δηλαδή αυτό ταμείο, είναι επειδή είναι μια πολύ καλή ιδέα, μια πολύ καλή μέθοδος για να μπορέσουν να επανέλθουν στο χρόνο απασχόλησης εκείνοι οι εργαζόμενοι που χρειάζονται αυτή την υποστηρίξη και δεν έχουν άλλες εναλλακτικέ δυνατότητες. Παραδείγματο χάνει. κλείνει ένα εργοστάσιο ή μεταφέρεται κάπου, δεν δίνει υποστήριξη σε όλους. Αυτό που σημαίνει όταν απολύεται κάποιος, το Ταμείο ρωτάει τι είδου κατάρτιση χρειάζεται αυτός ο ίδιος ο για να επανέλθει στον χώρο αποσχόλησης. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό δηλαδή αυτή η προσωπική προσέγγιση. Ο καθένα επιλέγει τι θεωρεί ότι χρειάζεται. Και είναι νομίζω πιο καλή αυτή η προσέγγιση από εκείνη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. με κάποια οριζόντια προγράμματα τα οποία τρέχουν σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος μέλος και ο σκοπός εκεί είναι να βελτιωθεί η κατάρτιση και των ενέργων και των ενεργών εργαζόμενων ε, για τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πρωτότυπο, διότι κατά τον τρόπο δίνεται η πρωτοβουλία στον άνεργο στο ποια διέξοδο θα διαλέξει για να βγει από την ανεργία. Οπότε βλέπουμε πόσο προοδευτικό είναι αυτό το ταμείο διότι προσαρμόζεται στις προσδοκίες αλλά και τις ανάγκες του εργαζόμενου. Πρόκειται για ένα ολόκληρο εργαστήριο και γι' αυτό και εμείς θα πρέπει αυτό να το αγκαλιάσουμε σαν ένα αυτόνομο ταμείο που υπάγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να επεκτείνουμε αυτές τις πρακτικές και στι υπόλοιπες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό δηλαδή να, να, να να, να μεταδοθεί το καλό και όχι οι κακέ συνήθειες του ΣΥΠΗΝ, αυτά που λειτουργούν λιγότερο καλά. και αυτό επομένως είναι η βασική, το, το, το ζουμί του αυτής της έκθεσης. Προσπαθούμε επομένως όλα αυτά να τα, να, να τα αποτυπώσουμε στην έκθεση. Αυτό είναι το πνεύμα που διαπνέει την έκθεση. Πώς επομένως όλα αυτά θα παγιωθούν, πώ θα βελτιωθούν Εδώ και ένα χρόνο έχει γίνει γνωστό ότι 200 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει το Ταμείο, ενώ, ενώ πριν από λίγο καιρό είχε μόνο 80. Πάντως οι, οι επιλέξιμοι έχουν αυξηθεί κατά 50% μέσα σε ένα χρόνο. Οι υποψηφιότητες έχουν τριπλασιαστεί 42 υποψηφιότητες ξέρω ότι είχαμε αυτή την τελευταία χρονιά. Σχεδόν μία υποψηφιότης εβδομαδίως. Επομένως βλέπετε ότι χρειάζεται να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό το ταμείο στο Ευρωκατημέλη γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα για το 2009 και το 2010. Πέραν αυτών. Βλέπετε ότι αρχίζει να βελτιώνει η λειτουργία. Από την άλλη μεριά έχουμε κάποια ε, στρεβλά φαινόμενα, κάποια, κάποιες, κάποιες αδιεξόδους. Έχουμε δηλαδή αυτά τα 50 πρόσωπα, 16 ψηφιότητες, οι 42 ε, ε, μέσα σε μια χρονιά που θα πρέπει να μελετηθούν, να αναλυθούν, χωρίς να κάτσουμε και να βρούμε έστω και έναν παραπάνω που να μπορεί να βοηθήσει για το προσωπικό. Επομένω άρχισαν τα στρεβλά, τα αρνητικά αποτελέσματα και γι' αυτό και κάποιες κυβερνήσεις άρχισαν να αμφισβητούν ε, αυτό το, τον οργανισμό, αυτό το ταμείο, ιδίως από πιο πλούσιες χώρες αυτό άρχισαν να λένε Πάντως σήμερα έχουμε ανέργους από πλούσιες χώρες και πλούσιες περιφέρειες οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για τις δράσεις του Ταμείου. Αυτό ακούγεται έτσι σαν παράδοξο. Όμως θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα βελτιωθεί η δραστηριότητα του Ταμείου. Αυτά και εν κατακλείδη έχω να σας πω για τις προτάσεις αυτές ότι θα πρέπει να τις υλοποιήσουμε σε τρεις φάσεις. Σε αμέσως επόμενες ε, εβδομάδες, μήνες θα πρέπει να δούμε τι διαδικασίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι μέσα στη διάθεσή μας, ούτω ώστε το ταμείο αυτό να γίνει πιο επιχειρησιακό, πιο λειτουργικό από πλευράς αυτού που είναι αυτός που θέλει τις υπηρεσίες του. Δηλαδή αυτός ο οποίος υπέστη μια ομαδική απόλυση. Αν λεφθεί απόψη τι δυνατότητες δίνονται από την Εθνική Νομοθεσία και τι μπορεί να γίνει από πλευράς ε, ε εθνική εργατική νομοθεσία, δηλαδή 12 με 16 μήνε που προβλέπονται όσον αφορά ε, την, ε, την όχληση, την προειδοποίηση για την απόλυση. Επομένως, είπαμε ότι το Ταμείο αυτό θα λειτουργεί μέχρι το 2011. Θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό, να δούμε πώς θα παραταθεί η λειτουργία του μέχρι το 2013, γιατί τότε λήγουν οι ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές. Θα πρέπει να βελτιωθεί ο σχετικό ασκονισμό. θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα κάνουμε μέσα από ένα χρονιά όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό αυτό το ταμείο. Επίσης, Πρέπει να σας πω ότι από το 2013 και μετά αυτό το ταμείο είναι δυνατόν να μπορεί να είναι εις θέση να έχει το δικό του προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν θα είναι τίτλος, αν θα είναι κονδύλιο, θα είναι πάντως ένα καθεαυτού ταμείο με αυτονομία. Είπαμε να είναι το παράδειγμα προς μίμηση αυτό για τα άλλα ταμεία και το κοινωνικό ταμείο και να μην κολλήσει τα δεινά, ας το πούμε έτσι, του κοινωνικού ταμείου, αυτά που δεν πάνε καλά. Θα πρόκειται επομένω για μια εξέλιξη, για ένα βήμα προόδου ιστορικό. Δεν είπα αυτό να το συζητήσουμε εδώ και τώρα. Θα πρέπει όμω να αρχίσει αυτή η προβληματική να αναπτύσσεται εν ώψη των επομένων δημοσιομικών προοπτικών. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν θα... Αν θα αρκέσουν αυτά τα, χρήματα που θα προέλθουν από τις εκριζώσεις του καπνού, τα 300 τόσα εκατομμύρια, θα δούμε. Αλλά πάντως ε, αυτό αργά και γρήγορα πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω και κλείνω ότι το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα τώρα είναι ότι μέσα σε αυτή την συγκυρία της οικονομικής κρίσης, κρίσης, μια που έχουμε τέτοια χτυπήματα τέτοια, που έχει δεχθεί η αγορά εργασίας, θα πρέπει να δούμε πώς δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση με ακόμα μεγαλύτερα χτυπήματα στην αγορά απασχόληση, αλλά πώς θα βοηθήσουμε τους εργαζόμενους στην Ευρώπη Πώς θα δείξουμε στους εργαζόμενους ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό τους. Άρα χρειάζεται αυτό το μήνυμα να στείλουμε. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθήσουμε μαζί με τις άλλες πολιτικές που τώρα ασκούμε ένα τέτοιο μήνυμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό ούτω ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την επαγγελματική ένταξη και την κατάρτιση. Και φυσικά να βοηθήσουμε και το κάθε κράτος μέλος να έχει αντίστοιχε καλύτερες, πιο αποτελεσματικέ στρατηγικές. Με αυτό το ταμείο. Ένα πραγματικό εργαστήρι. Ακριβώς γιατί δίνει προσοχή στο κάθε πρόσωπο χωριστά. Ευχαριστώ πολύ. Eh Ευχαριστώ τον εισηγητή. Έχουμε ανάμεσά μας και την κυρία Σαρτιέ από την άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία δίνομαι στο λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στη συζήτησή σας για αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εργαστήκαμε πολύ στο συγκεκριμένο θέμα μαζί με τον Μιγέλ Πόρτας. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθώ από τότε που τέθηκε η εφαρμογή η απόφαση του Συμβουλίου το 2007. Έχω δει πως εξελίχθηκε. Καταρχάς ίσχυσε κυρίως για τις επιχειρήσεις, αλλά μετά από την τροποποίηση του 2009 προσανατολίζεται στους εργαζομένους, όπως έλεγε ο κ. Πόρτας. Και εκεί έγκυται και η πρωτοτυπία του αν θέλετε. Αν πρέπει να υπογραμμίσω ε, κάποια συγκεκριμένα σημεία του ταμείου αυτού, είναι ότι απευθύνεται στους εργαζομένους, οι οποίοι δεν φύγονται μόνο από την παγκοσμιοποίηση αλλά και από την οικονομική κρίση με μαζικό τρόπο, σε έναν συγκεκριμένο τομέα, σε μια περιφέρεια, σε μια χώρα ή και σε δύο χώρες συνοριακά. Αυτό είναι το πρώτο, αν θέλετε, πρωτότυπο χαρακτηριστικό του. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του ταμείου αυτού είναι η μεγάλη ευελιξία που το χαρακτηρίζει. Εμείς θα θέλαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη και γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε στις συγκεκριμένε τροποποίησεις. Γιατί το λέω αυτό. Στα πλαίσια του τρόπου που εργαστήκαμε σήμερα, ιδιαίτερα στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Κοινωνικής Επιτροπής. Πήγαμε επιτόπου στην Ιρλανδία, είδαμε το τι συμβαίνει στο Λίμερικ, στους 2.500 απολυμμένους της επιχείρησης Dell. Εργαστήκαμε επίσης και με τους Γερμανούς και με τους Αυστριακούς για τον σωστό τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου ταμείου μέσω των ε, επιχειρήσεων, ε, μάλλον μέσω των συγκεκριμένων τρόπων μεταφοράς. Και βλέπει κανείς πως μέσα από το πρόγραμμα αυτό, από τη γνωμοδότηση την οποία συνέγρεψα για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η τοπική εμπειρία που έχουμε με τις επιχειρήσεις από τη Γερμανία και από την Αυστρία μας έδειξαν ότι απαιτούνται περαιτέρω τροπολογήσεις έτσι ώστε το ταμείο αυτό να είναι πιο χρήσιμο, πιο γρήγορο και πιο ευέλικτο. Οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στη γνωμοδότησή μου έχουν σαν στόχο θα έλεγα ε, μάλλον έχουν κατατεθεί από πέντε πολιτικές ομάδες. Δηλαδή βλέπουμε ότι στην Επιτροπή μου υπάρχει μια σχετική συνένεση η οποία έχει αρχίσει και διαφαίνεται ε, για τον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε το Ταμείο αυτό και αυτό νομίζω είναι συμβατό με την έκθεση του κυρίου Πόρτας. Πρόκειται για ένα ταμείο για το οποίο διαπιστώνουμε μια επιτάχυνση των αιτήσεων, της ζήτησης. Υπάρχει ταυτόχρονα και μια αύξηση των ποσών που θα πρέπει να χρειαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Αυτό που συναντά κανείς πολύ συχνά είναι ότι οι εργαζόμενοι που έχουν ανάγκη από το ταμείο αυτό είναι ότι είναι εργαζόμενοι που έχουν αρχίσει περίπου την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την απόλυση 20-25 χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία χωρίς καμία επαγγελματική συμπληρωματική επικύρωση, χωρίς επικύρωση των, της σταδιοδρομίας της επαγγελματικής τους και της απόκτησης επαγγελματικών ικανοτήτων. Αυτό είναι το μάθημα που παίρνουμε από τη λειτουργία του Ταμείου. Ότι δηλαδή ωφελώντας τους εργαζομένους θα πρέπει να επιτρέψει την επαγγελματική τους επανένταξη το ταχύτερο δυνατόν μέσω μιας εξατομίκευσης αν θέλετε των αναγκών. Ο λόγος για τον οποίο είναι ότι οι αποτυχίες τις οποίες συναντήσαμε όταν συναντώνται ακριβώς είναι ότι οφείλονται σε μια έλλειψη εξατομίκευσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα με συλλογικό τρόπο. Όταν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από μαζικές απολύσεις, πρέπει να δοθούν ατομικές αλλά και γρήγορες απαντήσεις. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ξεκινήσουν ε, διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Και θα πρέπει αυτή η διαβούλευση να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του ταμείου αυτού, ισχύω του ταμείου αυτού για την παγκοσμιοποίηση. Το τρίτο θέμα άπτεται των συμπερασμάτων του Μιγγέλ Πόρτας το ταμείο αυτό είναι χρήσιμο. Αλλά δεν μπορούμε συνεχώς να καλύπτουμε τις ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι λόγω της ανυπαρξίας πολιτικής κατάρτισης των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται, που δεν τους βοηθούν οι επιχειρήσεις αυτές να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητά τους. Πρέπει λοιπόν αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να λειτουργήσει σαν καταλήτης για να υπάρξουν αλλαγές θα πρέπει να μην είναι μόνο μεμονωμένο και εξατομικευμένο το ταμείο αυτό, αλλά να μπορεί να καλύψει και να προβλέψει κάποιες ε, μαζικές απολύσεις οι οποίες μπορεί ε, να υπάρξουν. Συμμετέχω σε αυτή την ομάδα που διαχειρίζεται λοιπόν το θέμα. Πρέπει οι διαδικασίες να απλοποιηθούν πρέπει να επιταχυνθούν να επιταχυνθεί η βοήθεια που δίδεται στους εργαζομένους από τη στιγμή που δημοσιοποιείται η απόλυση μέχρι τη στιγμή που έρχεται η βοήθεια πρέπει αυτοί οι ατελείωτοι μήνες που μεσολαβούν να μειωθούν. Φυσικά πρέπει να παραταθεί η ισχύ αυτού του ταμείου, είναι απαραίτητο αυτό γιατί βλέπουμε ότι η επιτάχυνση των αιτήσεων, η αύξηση των αιτήσεων αποδεικνύει ότι προστίθεται, σωρεύεται με την παγκοσμιοποίηση η οικονομική κρίση και έτσι αυτό το ταμείο καθίσταται ακόμα περισσότερο χρήσιμο. Να προσθέσω επίσης ότι θα πρέπει να δώσουμε στο Ταμείο αυτό μια μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα θα έλεγα. Ε, θα πρέπει να του δώσουμε μια καλύτερη θέση στην πολιτική μας και ο, ο προϋπολογισμός είναι ακριβώς αυτό το μέσο της πολιτικής που πρέπει να υπογραμμιστεί. Θα πρέπει να υπάρξει ένα ξεκάθαρο μήνυμα έτσι ώστε οι πολιτικές επαγγελματική ένταξη των πιο εύθραστων εργαζομένων να καλύπτουμε τις ανάγκες τους γιατί πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από το σχολείο χωρίς εκπαίδευση, χωρίς επαγγελματική κατάρτιση, χωρίς μαθητεία καν μερικές φορές και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα όταν μετά από πολλά χρόνια απολύονται. Πρόκειται για ένα χρήσιμο ταμείο, εν περιπτώσει, που βοηθάει για ένα καλύτερο ε, μέλλον του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ αγαπητέ Porteur et je me réjouis de la, la qualité de Ευχαριστώ του δύο συγκεκριτές μας και χαίρομαι για τη συνεργασία που διαγράφεται μεταξύ τη Επιτροπή ε, Προαπλογισμών και τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το τόσο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Οι δύο συγκριτέ μα που εργάστηκαν στενά συνεργαζόμενοι ε, κατέδειξαν ποια είναι τα προβλήματα. Αυτό το ταμείο έχει τώρα τρία χρόνια εμπειρία και είναι καιρό να έχουμε ένα πρώτο απολογισμό για να διορθωθεί ενδεχομένω κάτι, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες ε, διαδικασίε. Το θέμα λοιπόν, όπως μας υπενθύμησαν, είναι καταρχήν θα συνεχιστεί, θα διατηρηθεί το Ταμείο, προφανώς και οι δύο απαντούν θετικά Γνωρίζοντα όμω, όπως είπαμε, ότι αυτό το ταμείο προετοιμάστηκε για να βοηθήσει μάλλον τις επιχειρήσεις που ήταν θύματα του ανταγωνισμού, που σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση, και επίσης όχι απαραίτητο για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που είναι θύματα της κρίσης. Δεν είναι ακριβώ. το ίδιο. Και δεύτερον, τα κριτήρια που υπάρχουν για να ωφεληθεί κανένας από το ταμείο αυτό είναι τα σωστά κριτήρια. Είναι πολύ υπερβολικά ευέλικτα, υπερβολικά άκαμπτα ή τι. Και το τρίτο θέμα είναι η διαδικασία. Οι προθυμίε που ανέφερε ο κ. Χορτά είναι μακρέ. Έξι μήνε πριν ληφθεί μια απόφαση, 12 μήνε μεταξύ τη στιγμή που τα θύματα μιας μαζικής απόλυσης μπορούν να βρουν μια συγκεκριμένη λύση, θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα τμήμα της διαδικασίας που σχετίζεται με τις εσωτερικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Γιατί ακριβώς έχουμε μια πάρα πολύ βραδική διαδικασία, ότι μπορεί να κοινοποιηθεί δηλαδή μόνο το Ταμείο για κάποια συγκεκριμένη ε, κατάσταση, εφόσον υπάρχει μία απόφαση των ε, κοινωτικών οργάνων για την μεταφορά των πόρων αυτών. Προφανώ δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε μια κατάσταση στην οποία το Κοινοβούλιο διαχειρίζεται μια διοικητική διαδικασία. Στην αρχή ε, ελέγχουμε κάθε φάκελο, εντάξει, για να δούμε πώς λειτουργεί. Αυτό μπορούσαμε να τα κάνουμε όταν είχαμε λίγους φακέλους ε, κάθε εξάμεινο. Τώρα όμω που έχουμε λίγου φακέλου κάθε εβδομάδα, θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα διαχείριση. Προφανώ υπάρχει το πρόβλημα τη διαχείριση. Η... λύση ήταν αρκετά και ανατομική γιατί εγγράφεται το ένα ε, αριθμητικό στοιχείο χωρί να καλύπτει τίποτα από το στοιχείο αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό στην δημοσιονομική διαδικασία. Τώρα θα πρέπει να προσδιοθούμε βέβαια. ξέρω. έφτασε η στιγμή να προσδιοθούμε ή θα μπορούμε να παραμείνουμε ακόμα στα σύννεφα λίγο. Και μετά δείχνει το θέμα του μέλλοντος. Και εκεί το μήνυμα του εισηγητή είναι σαφές. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να διορθώσουμε την κατάσταση, να προσαρμόσουμε τη διαδικασία μέχρι το 2013 και μετά το 2013 με τις επόμενες δημοσιονομικές προβλέψεις θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα πιο εις βάθος. Εγώ έξω. Είμαι κάπως... Ε, ε, θα έλεγα ότι γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουμε δώσει τη δυνατότητα να διευκολυνθούν αυτοί οι εργασόμενοι μέσω του κοινωνικού ταμείου. Τι χρησιμεύει το κοινωνικό ταμείο αν δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Αν δεν το κάνει θα πρέπει να το κάνει. Οι παλιότεροι εδώ, τα θυμώντα, ότι στο παλιότερο καθεστώς των ιδιωτικών ταμείων υπήρχε ο στόχος 1, ο στόχος 2 και να, το 2β ή το 5β, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώς, που είχε σαν στόχο να βοηθήσει ακριβώς τις ζώνες που πλήττονται από την βιομηχανική αναπροσαρμογή. Ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν ε, χρηματοδοτείται πια από το Ιερωτικό Ταμείο. Κατά τη γνώμη λοιπόν αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να θέσουμε άμεσα πάνω στην έκθεση του κυρίου Πόρτας, αλλά θα πρέπει να το έχουμε κατά νου για τη σκέψη που θα κάνουμε για το μέλλον των περιφερειακών ε, πολιτικών συνοχής. Δεν είναι λογικό από τη μια μεριά να έχουμε έναν μηχανισμό πάρα πολύ πολύπλοκο που τον εισαγάγουμε κάθε 7 χρόνια, τον οποίο προβλέπουμε 40 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο και όταν ξαφνικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται από διεθνή ανταγωνισμό, από οικονομική κρίση, από αύξηση της υποκοσμιοποίησης, δεν έχουμε τίποτα σχέδια χέρια μας και αναγκαζόμαστε να βρούμε νέες διαδικασίες για να αφαιρέσουμε αυτά τα χρήματα από το κοινωνικό ταμείο και θα είναι εκεί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πάντα. θα πρέπει λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη μας ε, όσον αφορά τις ε, νέες δημοσιονομικές προβλέψεις και τις ε, κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές συνοχές. Τώρα έχουν ζητήσει μια σειρά μελών. Την λόγω κύριο Άγγλουντ κυρίω. Τσαγκαρο Δευτέρα είναι, να σας τα πω ή στα Σουηδικά. Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που έχουμε ένα δικό μας ηγητή και έχουμε και διάφορους σκιώδη συζητητέ. και εγώ σκιώδη συζητητή είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Υπάρχουν πολλά να πούμε εδώ και σα διαβεβαιώ ότι είχαμε πάρα πολύ έντονε συζητήσει στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Γιατί όταν κάποιο πλήττεται από την παγκοσμιοποίηση, ο στόχο ήταν να βοηθεί από το ταμείο. Τώρα βέβαια η κατάσταση έχει αλλάξει πάρα πολύ σημαντικά. Ο σημερινό στόχο είναι διαφορετικό από τον αρχικό. Και θέλω να σας πω ότι στη δική μας πολιτική ομάδα, στους φιλελεύθερους, υπάρχουν πάρα πολλές κριτικές. Ίσως αυτό ισχύει και για άλλες πολιτικές ομάδες και γι' αυτό θα ήταν καλό ίσως γενικά να αξιολογήσουμε αυτό το ταμείο και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε το ταμείο αυτό στο μέλλον. Εκτός αυτό θα ήθελα να σας πω ότι καταρχήν θεωρώ ότι δεν είναι θέμα του δημοσίου τομέα, να αναμειγνύεται σε αυτά τα θέματα. Δεν μου αρέσει λοιπόν και πολύ η ιδέα, αλλά εντάξει. Άπαξ και έχουμε το τομέα θα πρέπει να φροντίσουμε να λειτουργεί σωστά. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμή ήταν κάπως τυχαία θα έλεγα. Μπορούμε να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ε, ε, καταβάλουν τα χρήματα δεν ήταν πάρα πολύ καλά μελετημένος, ήταν μάλλον τυχαίο εξαρτάται από το ποιος δρούσε εκεί, ποιο είχε ζητήσει περισσότερα. Ε, δεν μου φαίνεται και αυτό πάρα πολύ καλό, εδώ που τα λέμε. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ε, πώς θα προσανατολιστεί το ταμείο στο μέλλον. Εκτός αυτού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηρές οριακές τιμές. Ε, πληρωμή των χρημάτων είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Μόνο όταν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη αριθμοί απολυμμένων εργαζομένων κλπ. Αλλά υπάρχει και το θέμα των μεμονωμένων τραγωδιών. Δηλαδή το θέμα δεν είναι πόσοι απολύονται, αλλά το θέμα είναι πόσο πλήγεται ο καθένας από την απόλυση αυτή. Και γι' αυτό νομίζω ότι στην Επιτροπή ε, Οικονομικών Υποθέσεων θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε σε ένα κείμενο και να έχετε μια επικοδοματική τοποθέτηση της Επιτροπής αυτής. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσα πραγματικά να πω ότι αυτό το Ταμείο θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω. Είναι εξελιχθεί ή να καταργηθεί. Γιατί εδώ θα πρέπει να εξηγάμε προς πολίτες γιατί έχουμε αυτό το ταμείο έτσι, γιατί εάν θέλουμε να αιτιολογήσουμε το ταμείο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί δίκαιο σε όλη την Ευρώπη. Είμαι λοιπόν εγώ υπέρ μια επικοδομητική κριτική συζήτηση να έχουμε καλά τελικά αποτελέσματα. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Ο Σαλβατόρ έχει το λόγο. Ακριβώ, Πρόεδρε, επειδή θέλουμε να σημειώσει προόδους το Ταμείο. Γι' αυτό και θέλουμε να το μεταρρυθμίσουμε και γι' αυτό κάθισε ο συνέδελφος Πόρτα και έγραψε αυτή την εκθέση τη πρωτοβουλία για την οποία τον συγχαίρουμε Όλε οι πολιτικέ πτέρυγε του Κοινοβουλίου, μια που είναι πολύ χρήσιμα τα όσα προτείνει. Βοηθάει τη συζήτηση, έγινε και διαβούλευση από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστούμε πραγματικά. Και θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε τι πρώτε αντιδράσει ε, όπως διατυπώθηκαν των πολιτικών ομάδων και επί τη βάση αυτών κάθισε και έγραψε αυτή την συνενετική έκθεση. Οπότε συγχαρητήρια για τον ε, τόσο νεωτερικό τρόπο με τον οποίο δούλεψε. Πάρα πολύ παράδοξη είναι τώρα η, να πούμε, η κατάσταση. Ε, είναι πάρα πολύ ιδιόμορφη η φύση αυτού του ταμείου γιατί οι δημοσιογικές προοπτικές δεν έλαβε υπόψη το Συμβούλιο αυτό το ταμείο αλλά ούτε και το Κοινοβούλιο το σκέφτηκε μια που θεώρησε ότι πάντα αυτό το ταμείο θα είναι κάτι το περαστικό, το σημειακό και έτσι θα πληρώνονταν όλε οι σχετικέ ενέργειε από το Κοινωνικό Ταμείο. Έχουμε μόνο μια κατάσταση ανάγκε για εργαζόμενου και για επιχειρήσει. Έχουμε προβλήματα τη παγκοσμιοποίηση. Έχουμε τα προβλήματα των εργαζόμενων από την οικονομική κρίση. Για όλα αυτά προβληματίζομαι και έχω μια απορία και αβεβαιότητα. Πώς θα γίνει με αυτή την ανεργία που έχουμε στα 27 κράτη-μέλη να έχουμε αιτήσει και ανάγκες από όλους. Για μια πολύ λέει ότι δεν προέρχονται από όλους οι αιτήσει βοηθείας, αλλά μόνο από τα πιο πλούσια κράτη. Αυτό πρέπει να κάτσουμε και να το δούμε. Δεν θα υπάρχει κάποιος λόγος, δεν μπορεί. Γιατί κάποια κρατημέλη έχουν ε, ανεργία σημαντική και δεν προσφεύγουν στο ταμείο. Πάντως, όπως λέει ο συνάδελφος Πόρτας, προσέχει τον καθένα χωριστά. Εξατομικευμένο είναι το έργο του ταμείου αυτού, το οποίο νομίζω ότι προσυδειάζει στη φύση ενό διασωτικού ταμείου. Η πολιτική μας ομάδα θέλει να μην έχει αυτό το Ταμείο Προξενοποίησης χαρακτήρα διαρθρωτικού ταμείου. Εδώ επομένω υπάρχει διαφωνία. Να κάτσουμε και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το ταμείο και αυτό το συστήσουμε όταν κάτσουμε και συστήσουμε το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Θα κάτσουμε όμως και θα αναλύσουμε και θα αποφασίσουμε το αν θα ισχύσει και πόσο επικουρικότητα στην κοινωνική πολιτική. Να έχουμε μια κοινωνική πολιτική αυθεντικά κοινωνική. Αυτό θέλουμε. Όμως από την άλλη μεριά <clears throat> βρίσκουμε μπροστά μας το το κάνουμε αυτό την επικουρικότητα. Να μην δούμε σαν κομμάτι του, της διαρθρωτικής πολιτικής αυτό το ταμείο, να το δούμε σαν με ένα παρακλάδι, μια φυσική εξέλιξη του Γενικού Ταμείου, ε, το οποίο από πλευράς οικονομικής κρίσης δεν έχει πετύχει και πολλά πράγματα. Να κάτσουμε πώς να κάνουμε αυτή την ανάλυση όταν έρθει η ώρα για να αποφασίσουμε εμείς εδώ σε ποια πλαίσια στο μέλλον θα κινηθεί αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, αυτήν που θέλουμε να ασκήσουμε. Πώς νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένη η συνταγή που χρησιμοποιήθηκε. Και νομίζω ότι υποκρύπτει κινδύνους το να κάτσουμε και να θεωρήσουμε ότι αυτό το ταμείο είναι κομμάτι του, των διαθωτικών ταμείων, κύριε Πόρτα. Α τα αφήσουμε αυτό και όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε στο μέλλον διαπραγματεύσει, τότε να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά τι ε, τροπολογίε, νομίζω ότι ο συνάδελφος που έχει αναλάβει πρόκειται να σας πει τη γνώμη του για την κάθε μία τροπολογία χωριστά. Ευχαριστούμε Σαλβαδόρ, λέει ο πρόεδρος και δίνει το λόγο στην κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή και συγχαρητήρια. Πρόκειται για αυτό το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Όντω είναι πρωτότυπο αυτό το ταμείο. Τα σημεία ασφυξία έχουν επισημανθεί, τα καλά και τα κακά, τα είπε και ο πρόεδρο Λαμασούρ, τα είπε και ο διασυνονιστή μα, ο κύριο Γκαρίγα. Θέλουμε να αποκτήσει όμως διαρκή χαρακτήρα αυτό το ταμείο και να έχει το δικό του προπολογισμό. Και ως το είπε δεν μας νοιάζει όπου έρχονται τα χρήματα οι πρικότητες του ταμείου. Σωστό όμως ε, τελικά το μέλλον του θα εξαρτηθεί από το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Οι διαφορές είναι οι εξής, ότι δεν έχουμε εξατομικευμένη ε, κατάρτισε και την άλλη μεριά ότι διαφέρουν οι καλυπτόμενες περιοχές σε σχέση με το κάθε ταμείο. Είπαμε ότι το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης ασχολείται κυρίως με τις πιο πλούσιες περιοχές και χώρες. Έτσι, να δούμε τι γίνεται τι τρόποι χρηματοδότηση υπάρχουν πέραν του κοινωνικού ταμείου. Πώς δηλαδή μπορούμε να κατευθύνουμε σε περιοχές που δεν είναι περιοχές συνοχής κάποιους πόρους από το Ταμείο Συνοχής. Συμφωνώ για τη μείωση του χρόνου. και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δούμε τι ε, λύσεις μπορούμε να αναζητήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την, την εξάλληψη των ε, ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων. Ακριβώς όπως ε, αναφέρεται έχουμε 500 ευρώ με 22.000 ευρώ διαφορά. Είναι ένα προς, προς, προς 40 η αναλογία της, της ανισότητας. Είναι δηλαδή τρομερό. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι άλλο τώρα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο είναι το ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες της ε, Ένωσης δεν συμμετέχουν στο Ταμείο και έχουν πρόβλημα ανεργίας. Ποιος είναι ο λόγος. Είναι με μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση του κοινωνικού ταμείου. Είναι γιατί ίσως είναι πιο απλό το να προσφεύγει κανείς στο κοινωνικό ταμείο. Να το μελετήσουμε, να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Να δούμε σε τι υπερτερεί αυτό το ταμείο σε σχέση με το κοινωνικό ταμείο και αντιστρόφως. Είπαμε για την εξατομικευμένη κατάρτιση, είπαμε ότι πρόκειται για πραγματικό εργαστήρι κατάρτισης, αλλά και όσον αφορά την ε, παιδεία και όσον αφορά την κατάρτιση της εξοδομικευμένας και το ένα και το άλλο είναι δύσκολα πράγματα. Ε, χρειάζονται συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τι έχουμε αποσπάσει εδώ από αυτή την υπόθεση της εξοδομικευμένης κατάρτισης. Εδώ τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Κομισιόν, αλλά όχι αυτό το τι ακριβώς πετύχαμε. Αυτό πρέπει να μας πει η Κομισιόν να κάτσει η Κομισιόν και να δει αυτού, οι νέες μορφές κατάρτισης πόσο ωφελήσει. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Αν πρέπει να δούμε ότι είχε κοινωνική λειτουργία αυτός ο μηχανισμός διότι έχει παράσχει σε χώρες που δεν είναι χώρες συνοχής κάποια στήριξη πάντως όλες οι χώρες είναι ίσες και ακούσαμε την εμπειρία της Λιθουανίας στην ακρόασή μας Πρώτη μια χώρα που είναι από τις πρώτες που καλύφθηκε από αυτόν τον μηχανισμό και αν θέλουμε να κάτσουμε και να συγκρίνουμε αυτό το ταμείο με το κοινωνικό ταμείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ότι το Γενικό Ταμείο είναι το νοσοκομείο, είναι ο γιατρός της πόλης για την ε, πρόληψη, για την ιατρική αγωγή, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση είναι τα, τα κατεπήγοντα περιστατικά που ασχολείται με τα πάρα πολύ σοβαρά ατυχήματα, σώζει ζωές και κατόπιν έρχεται η, ιατρική τακτική αγωγή. Άρα να μην καθόμαστε και να υποτιμούμε το ένα ή το άλλο. Καλή είναι και η υπηρεσία των κατεπηγόντων, αλλά... Κύριε Μποκρός, έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ επιφυλάσσομαι πολύ περισσότερο για αυτό το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης πολύ περισσότερο από όσο προλαλήσαν οι συνάδελφοι. Διότι, κατά τη γνώμη μου, η αλλαγή των κανόνων του παιχνιδιού δεν λέει για με πολλά πράγματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Επίσης, θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε πόσα χρήματα έχουν ε, μείνει αναξιοποιητά. Πόσα κονδύλια μείνει αναξιοποιητά γιατί και αυτό έχει να κάνει με την επιτυχία στην πράξη. Γιατί στην αρχή θεωρήθηκε ότι ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργούσε και ότι θα έπρεπε να γίνει προσαρμογή αυτού του μηχανισμού και τελικά έγινε η προκάτωση πιο μεγάλη. Όμως η συνέπεια είναι ότι κάνει τώρα πιο πολλά πράγματα, αλλά δεν πιο αποτελεσματικό. Άλλο λοιπόν η, η απόδοση και άλλο η αποτελεσματικότητα. Και οι προηγούμενοι, οι αγορητές που πρέπει να αποφύγουμε, την κατάσταση κατά την οποία αυτό το ταμείο θα καταλήξει ένα διαρθωτικό ταμείο για τις πιο πλούσιες χώρες. Ήδη είναι κάτι τέτοιο, άρα αργά. Πολύ αργά τα λέτε αυτά αλλά υπάρχει και ένα τελευταίο και πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αφορά κάποιες ε, εταιρείε οι οποίες αποφασίζουν την επανεγκατάσταση. Γνωρίζουν την ύπαρξη του Ταμείου και άρα είναι ακόμη πιο σημαντικό να λαμβάνεται αυτή η απόφαση γιατί ένα μεγάλο σημαντικό ποσό των δαπανών μπορεί να μετακυλιστεί στην Ευρώπη σαν κοινωνική ενίσχυση. Επομένως αυτό είναι στρεβλή εκδήλωση του καπιταλισμού. Ακόμα και αν γίνεται αυτή η μεταφορά από στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και ή ακόμη αν πηγαίνει αυτή η επιχείρηση καπ' αλλού επομένως. Το τελευταίο πρόβλημα το οποίο κάποιοι ανέφεραν, κάποια σκληρά συμπεράσματα, είναι ότι εδώ υπάρχει επικάλυψη σε σχέση με άλλα μέσα πολιτικής τα οποία ισχύουν. Δυστυχώς έφυγε η συγκεκριμένη κυρία Αντρεγεύσκα, όμως θα ήθελα, όπως είπε και ο Τζιμ, είναι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως στη ακρόαση. πώς θα αναδιαρθρώσουμε τον προπολογισμό και πώς θα μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε εκείνα τα όργανα, τα μέσα πολιτικής τα οποία είναι τα πιο σημαντικά για να μπορούμε να έχουμε σύνδεση πιο στενή της κατάρτιση, της παιδείας με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης να πετύχουμε πάλι σωστή απασχόληση, να μην καθόμαστε να έχουμε κατάτμιση τόσα διαφορετικά όργανα και εργαλεία που το ένα σχεδόν με το άλλο. Να ένα καλό παράδειγμα. Μπορούμε αυτούς τους πώς να τους χρησιμοποιήσουμε τόσο ώστε να ενισχύσουμε, παγιώσουμε τα υπάρχοντα όργανα, ιδρύματα που τα ανέφερε στην της κ. και μπορεί να πετύχει τους σκοπούς του το ταμείο αυτό ακόμα καλύτερα. Παρά το να χρειαζόμαστε για να φτιάχνουμε χωριστά όργανα αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ συνάδελφε, θέσατε πολλά θέματα. Ιδιαίτερα το λεγόμενο θέμα του moral hazard. Κάθε φορά που υπάρχει ένα σύστημα βοήθειας προς κάποιον που έχει δυσκολίες, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι ένα κράτος, ένα κράτος μέλος της Ένωσης, της ζώνης ευρώ ή και εκτός ζώνης. Και Λαβία, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω κάποιες πλευρές της συζήτησης που ίσως να μην υπογραμμίστηκαν ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Το πρώτο είναι ότι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται από αυτό το χρηματοδοτικό μέσο είναι 17 από τις 27 χώρες. Αυτό είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα μετά από την τροποποίηση του ταμείου αυτού που καλύπτει και τις ανάγκες των εργαζομένων. Η κρίση έχει χτυπήσει όλη την Ευρώπη όμως και όχι μόνο ορισμένες χώρες. Τίθεται λοιπόν το θέμα, το ταμείο αυτό, το μέσο αυτό είναι γνωστό στην Ευρώπη. Και ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρώπης οι ίδιες προϋποθέσεις για τη χρήση του μέσου. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο σημειώθηκε από πολλούς, είναι το πρόβλημα της κατανομής των παρεμβάσεων ανάμεσα σε αυτές που καλύπτονται από το κοινωνικό ταμείο και όχι. Και στο εσωτερικό του κοινωνικού ταμείου υπάρχουν δυνατότητες για την ανταγωνιστική θα έλεγα ικανότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της επιχείρησης. Αντίθετα, το κοινωνικό μέσο, το κοινωνικό ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματά του για να εκπαιδεύσει εξ αρχής τους εργαζομένους που είναι εκτός εργασίας και να τους εντάξει. Το θέμα είναι βέβαια ότι πρέπει να είμαστε εδώ κάπως προσεκτικοί. Θα πρέπει εμείς το κοινωνικό ταμείο να το χρησιμοποιήσουμε βελτιώνοντάς το. Επειδή δεν είναι το πιο κατάλληλο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το απομακρύνουμε εμείς εντελώς. Θα πρέπει εμείς να χρησιμοποιήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού ταμείου που θα επιτρέψουν, θα επιτρέψουν την επαγγελματική επανένταξη των εργαζομένων. Αυτών που είναι εκτός βέβαια εργασίας ουσιαστικά Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δυνατότητες χρήσης ε, και του καινούριου μέσου ε, που καλύπτουν τους εργαζομένους. Στο παρελθόν δεν υπήρχε ομοιογένεια στις παρεμβάσεις του Ταμείου ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Είναι σαφές ότι κάποιοι πιο συγκεκριμένοι κανόνες για τη λειτουργία του Ταμείου αυτού είναι απαραίτητοι, έτσι ώστε όταν υπάρχει κακή χρήση των μέσων αυτό να διορθώνεται. Απ' την άλλη θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όλα τα μέσα τα οποία έχουν σαν στόχο και όλες οι διαδικασίες που έχουν επίσης σαν στόχο την μείωση του χρόνου παρέμβασης, του χρόνου κινητοποίησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να επιδιωχθούν έχουμε να κάνουμε με ένα μέσο το οποίο καλύπτει έκτακτες καταστάσεις. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μειώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον χρόνο που μεσολαβεί. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν τις βελτιώσεις τις οποίες προτείνει ο κύριος Πόρτας. Μία τελευταία πλευρά που πρέπει να υπογραμμίσω αφορά τον χρόνο ακριβώς, το να παραταθεί η δράση του ταμείου αυτού μέχρι το τέλος αυτής της προγραμματικής περίοδου, μέχρι το 2013 είναι χρήσιμο. Το να το μετατρέψουμε σε κάτι το διαφορετικό όμως δεν νομίζω ότι είναι επίκαιρο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμο με αφορμή τις διαπραγματεύσεις για τις νέες δημοσιονομικές τρόπικες. να επανεξετάσουμε τον ρόλο του κοινωνικού ταμείου και να επανεντάξουμε σε αυτό κάποιες από τις δραστηριότητες που έχει σήμερα το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση, ιδιαίτερα σε μια εποχή τόσο δύσκολη και απαιτητική όπως η σημερινή. Τρούπελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κοιτάξουμε τα πλανεκτήματα και τα ανεμοκτήματα αυτού του μέσου του Ταμείου Αποφύγησης τη Προγραμματίσης. Δημιουργήθηκε από τους ηγέτες Ευρώπης σαν ένα μηχανισμό παρέμβασης και τους έδωσε μια πολιτική ορατότητα. Ήταν το μωρό, αν θέλετε, του Μπαρόζο. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι είναι τμήμα του συνόλου της, ε, του πολιτικού παιχνιδιού. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή το θεωρώ σαν ένα πολιτικό μέσο του τέλους ε, της ε, διαδρομής, θα πρέπει να εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε με τη Συντόνια αν θέλουμε να αλλάξει η άποψη όσον αφορά την εκπαίδευση και όλη την έννοια της εκπαίδευσης αυτής μέσα στα πλαίσια του επιστημονικού προγράμματος και του προγράμματος του 2020 θα πρέπει να δούμε ότι είναι πιο σημαντικό να επενδύσουμε σε μαθητές, σε φοιτητές για στη διαβίου μάθηση και όχι να καταλήξουμε μόνο σε αυτό το πολιτικό μέσο που είναι το έσχατο μέσο κατά κάποιον τρόπο. Γιατί νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να δράσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και ακόμα και αν υπάρχουν λοιπόν επιχειρήματα ορατότητας υπάρχουν καλά επιχειρήματα που λένε ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε κάποιες συγκεκριμένε περιόδους του χρόνου ή της συγκυρίας και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα διαφορετικά ταμεία και τις πολιτικές παιδείας για να είναι ξεκάθαρη η προσέγγιση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να επενδύσει περισσότερο και να συγκεντρώσει προσοχή στο θέμα των μελλοντικών επενδύσεων. θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τα μειονεκτήματα, θα πρέπει να μάθουμε ποια είναι τα πραγματικά πλεονεκτήματα και να έχουμε ένα συνδυασμό διαστατικών ταμείων και διαβίου μάθησης. Ευχαριστώ, Έλγα. Ο κύριος Ντάρτεν. Για τη σοσιαλιστική ομάδα <clears throat> θα πω ότι συμφωνούμε πολύ με τις προτάσεις του κυρίου Πόρτας. Είχαμε την ευκαιρία να το το εκφράσουμε. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι κάνατε μια σωστή παρουσίαση του προβλήματος και το βασικό πρόβλημα που είναι η διατήρηση ή μη στο μέλλον του μέσου αυτού. Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το μέσο αυτό έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα την εξατομήκευση των τρόπων εφαρμογής του. Έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, έχει μεταρρυθμιστεί εδώ και λίγους μήνες και διαπιστώνουμε ότι είναι όλο και πιο επιτυχές. Κρίμα βέβαια που υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή του μέσου αυτού, αλλά αυτή είναι η διαπίστωση την οποία κάνουμε. Νομίζω ότι η χρησιμότητα ενός τέτοιου μέσου και το βαφτίζουμε όπως θέλουμε, ξέρετε, το μέσο αυτό. Το συμπεριλαμβάνουμε στο κοινωνικό ή δεν το συμπεριλαμβάνουμε στο κοινωνικό, το τροφοδοτούμε με διαφορετικούς τρόπους, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Νομίζω όμως ότι η μεταφορά την οποία είπατε έχει νόημα. Και νομίζω ότι η παρομοίωση μάλλον που κάνατε με, τα νοσοκομιακές, με τις νοσοκομιακές επιχειρήσεις είναι αληθινή. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν ανάγκες νοσοκομιακές, δυστυχώς απ' την άλλη. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί. Είναι τέλειο το ταμείο αυτό, όχι βέβαια. Τέλειο δεν είναι. Η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί, να εκλεπτυνθεί η παρέμβασή του, η δυνατότητα παρέμβασης που έχει θα πρέπει να καταστεί προσβασιμότερο ιδιαίτερα στις περιφέρειες όπου ο κοινωνικός ιστός επικαλύπτεται από έναν ιστό επιχειρήσεων ο οποίος είναι κυρίως μικρού και μικρότερου μεγέθους. Είναι κατεπίγουσα η βοήθεια την οποία δίδει και γι' αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από ε, ταχύτητα παρέμβασης. Αυτό το κάνει και ο εισηγητής μας στον τομέα της απασχόλησης. Πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Θα πρέπει επίσης να εμπλακούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικοί εταίροι λόγω ακριβώς των χαρακτηριστικών αυτής της βοήθειας που θα πρέπει να είναι όπως είπαμε εξατομικευμένη θα πρέπει όλοι οι εταίροι οι οποίοι γνωρίζουν τις ανάγκες επιτόπου που βιώνουν την επιχείρηση και τον κόσμο της εργασίας να συμμετέχουν το ταχύτερο δυνατόν να προλαμβάνουν εν πολλής κάποιες κρίσεις. Σε επίπεδο λοιπόν εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και γι' αυτό η σοσιαλιστική ομάδα μέσω των τροπολογιών της θα συνεισφέρει στην επεξεργασία του κειμένου του εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Σούριαν. Στα Ουγγρικά. Ακό. Ακούω αυτά τα οποία συζητούμε και μου δημιουργεί την εντύπωση ότι η Επιτροπή μας αποδεικνύει ότι δεν ασχολούμεθα μόνο με το του προπολογισμού αλλά και με τα ταμεία και τη χρήση τους. Μου δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτή η τόσο πλούσια συζήτηση. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία με τα οποία δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ για το ότι ο κίνδυνος είναι να μην μπορούν να έχουν προσβασιμότητα επιχειρήσεις στο ταμείο. Για την γνώμη μου δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πάνε σε πηγές αυτά τα χρήματα, ούτε μια δεκάρα. Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, όλα αυτά τα χρήματα τα <clears throat> καταβάλουν στους ε, απολυθέντες, τους άνεργους, στους εργαζόμενους. Όμως, ανακύπτει το εξής ερώτημα. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χειριστεί αυτό το πρόβλημα γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ευρώπης οι απολύσεις. Και οι άνεργοι. Είναι καθήκον το να ασχοληθούν με αυτούς τα κράτη-μέλη. Όπως ο έχουμε ομαδικές απολύσεις θα πρέπει να εκταμιεύονται πόροι για την κάλυψή τους. Άρα θα πρέπει να κεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί που είναι πιο σημαντικό το ενεργήσει η Ένωση παρά τα κράτη-μέλη. Φυσικά σε κάποιες περιπτώσει μπορεί να κρυθεί ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει τότε αυτό το ταμείο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το, το του. μπορούσαμε να πούμε, αντί για αυτό το ταμείο, Μήπω θα μπορούσαμε με άλλο τρόπο να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Με εκατοντάδε εκατομμύριων ευρώ για να ασκήσουν τις πολιτικές που χρειάζονται. Ξέρετε με έναν Φινλανδό συνάδελφο, ταξιδέψαμε στη χώρα του, πήγαμε σε ένα εργοστάσιο και Κατά αυτή μας την επίσκεψη διαπιστώσαμε ότι εκεί έχει κάνει δουλειά. Έχει επιτελέσει έργο αυτό το Ταμείο της ε, Παγκοσμιοποίησης. Βρισκόμαστε στη μέση της διαδρομής ε, των δημοσιογών προοπτικών. Έχουμε αυτά τα αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ θα τα κινητοποιήσουμε μέσω κάποιων εμβασμάτων μεταφοράς πόρων. Θα πρέπει επομένω να δούμε πώς θα αλλάξουμε την μεθοδολογία της εργασίας μας και να δούμε πώς στις δημιουργικές προοπτικές θα μπορέσουμε να καλύψουμε τους πόρους που πρέπει να κινητοποιηθούν. Αυτό είναι το ερώτημα. Προσωπικά προτιμώ να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το ταμείο και κατά τις επόμενες δημοσιογικές προοπτικές, αλλά ίσως κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Άρα θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας μας. Ακούσαμε τα υπέρ και τα κατά. για την ένταξη και αυτού του ταμείου στην προσπάθεια κινητοποίησης πόρων για το Γενικό Ταμείο. Αν όμως έχουμε κάποιο είδου αιτήσει μεταφοράς πόρων, τότε χρειάζεται διορθωτικό προϋπολογισμός. Ίσως τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά πώς. Δηλαδή, πρέπει να κινητοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε την σημερινή, την ισχύουσα νομική βάση. Ελπίζω ότι θα βρει η Επιτροπή μας τη λύση. Το πώς θα εξευρεθούν οι πόροι που χρειάζονται. Τα ποσά που χρειάζονται. Αυτό να σκεφτούμε. Και θα πρέπει με κάθε τίμημα να συνεχίσουν να υπάρχουν τα κονδύλια τα οποία ήδη προβλέπονται. να σκεφτούμε. Μας μένουν κάποιες εβδομάδες πριν την ε, τέταρτη μεταρρύθμιση. Να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε κάποιους πόρους που δεν το εκμεταλλευτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να μια λύση. Έτσι νομίζω έχουν τα πράγματα σήμερα και πάντως θα πρέπει να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Νομίζω ότι οι προτάσει του έφεραν κάποιε φρέσκε ιδέε, τροφοδότησαν τον προβληματισμό μα και έχουμε και κάποιε τροπολογίε ευχαριστώ. ευχαριστώ, Ιγκε Gressler. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω και η κυρία Τρόπερ, θα ήθελα να αναφερθώ στην επίδειξη του Ταμείου αυτού και ότι αυτό που θέλαμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε χρήματα που δεν είχαμε δαπανίσει. Αυτό ήταν ο στόχο μα δαπανίσουμε τα χρήματα που είχαμε περισσέψει στο προπλησμό. Τώρα δαπανούμε χρήματα που δεν έχουμε. Αντιστρέφουμε τελείω δηλαδή την κατάσταση. Και νομίζω ότι εάν δεν αφιερώσουμε καλύτερα τα υπάρχοντα ταμεία, ανάλογα με τους στόχου που έχουμε αυτή τη στιγμή, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Δηλαδή με τους, ε, τα παλιά ταμεία χρηματοδοτούμε ορχιδέες θα έλεγα, δηλαδή πράγματα που δεν χρειαζόμαστε κατά βάση. Και έχουμε τώρα νέα ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει. Θα πρέπει λοιπόν να μην δώσουμε εσφαλμένα κίνητρα. Υπάρχει ένα έλεγχο από την ε, Διεθνή Τράπεζα που λέγεται Doing Business και σύμφωνα με την σειρά αυτή η Ελλάδα είναι στη θέση 109. Άλλε χώρες που παίρνουν χρήματα από το ταμείο αυτό πάλι δεν έχουν καλή θέση. Και θα ήθελα να σας πω ότι η Ρουάντα είναι στη θέση 67. Θα πρέπει δηλαδή να επιβραβεύουμε εκείνες τις χώρες που δεν δημιουργούν ιδανικές προποθέσει για την οικονομία. Να δώσουμε κίνητρα για την καλή διαχείριση, τις καλές επιχειρήσεις. θέλουμε να έχουμε μια ε, καλύτερη ε, αντιμετώπιση γιατί εδώ χρηματοδοτούμε ε, καταστήσεις οι οποίες οπωσδήποτε δεν θέλουμε να διονυστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Τελευταίος ο μιλητής. Μπάρμπαρα Ματέα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα με καθυστέρηση. Δεν μπόρεσα να ακούσω διαζώντος τον κύριο Πόρτερ Σχετικά με τις ομιλίες τις οποίες παρακολούθησα, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για τη χρησιμότητα του συγκεκριμένου μέσου. Όπως είπε η κυρία Τρούπελ, το ταμείο αυτό γεννήθηκε από μια ιδέα, θα έλεγα, μετά από μια πρωτοβουλία πολιτική του Επιτρόπου Μπαρόσο. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά συζητάμε τη σημασία του ταμείου αυτού, του μέσου αυτού σήμερα. Άσχετο λοιπόν για τον λόγο με τον οποίο δημιουργήθηκε, έχει σημασία το μέσο αυτό και θα πρέπει να δούμε τη χρησιμότητά του και αν υπάρχει ανάγκη για τη διατήρηση του συγκεκριμένου ταμείου και εγώ πιστεύω ότι είναι χρήσιμο το ταμείο αυτό και δεν συζητάμε μόνο την κατάργησή του. Συγχαίρω τον κύριο Πόρτας, έχει κάνει μια λεπτομερή παρουσίαση των δυνατοτήτων του ταμείου αυτού, του μέσου αυτού. Η ανάλυση του συγκεκριμένου ταμείου δείχνει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τη χρήση του συγκεκριμένου ταμείου. Για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε λοιπόν, Ποιες από τις ιδέες που ακούστηκαν θεωρώ ότι είναι οι πιο χρήσιμες. Θα ήθελα να αναλύσω μαζί σας κάποια σημαντικά σημεία. Για την παράγραφο 5 θα συμφωνήσουμε όλοι, να γίνουν δηλαδή οι διαδικασίες πιο γρήγορες. Από το αίτημα του κράτους μέλους μέχρι την λειτουργία του ίδιου του Ταμείου. Υπάρχουν και άλλες ιδέες όμως χρήσιμες. Οι αιτήσει θα πρέπει να προπαρασκευαστούν από τα κράτη-μέλη τη στιγμή που ανακοινώνεται η ομαδική απόλυση και όχι τη στιγμή που γίνεται γεγονός και θα πρέπει επίσης να μπορούν να κατατίθενται στην γλώσσα του κάθε κράτους μέλους και όχι σε μία από τις γλώσσες εργασίας. Θα πρέπει να ενισχυθεί το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τις αιτήσει αυτές. Και ο εισηγητής αναφέρθηκε και στον χρόνο σεβασμού των 15 που απαιτείται για την περίοδο κινητοποίησης και την πληρωμή φυσικά και είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τον χρόνο ανάλυσης των αιτημάτων αυτών. Η ανάλυση ουσιαστικά γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 μήνες μετά την κατάθεσή τους και αυτό είναι απαράδεκτο. Για την παράγραφο 6 είμαι υπέρ φυσικά του να εξεταστούν τα αιτήματα που έχουν ε, φτάσει στην Ολομέλεια και επίσης και να αντιμετωπιστούν ομαδικά θα έλεγα οι συλλογικές περιπτώσεις απολύσεων. Φυσικά γνωρίζω ποια είναι η δημοσιονομική επικαιρότητα θα έλεγα, αλλά παρόλα αυτά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να ελέγχουν την διαδικασία για την κινητοποίηση του συγκεκριμένου ταμείου. Για την παράγραφο 8, και θα συμφωνήσουν πολλοί συνάδελφοι μαζί μου, να παραταθεί δηλαδή το χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης από το 11 μέχρι το 13. Και δεν είμαι υπέρ ε, της αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 55% γιατί αυτό ουσιαστικά θα μειώσει την διαφορά ανάμεσα στο κοινωνικό ταμείο και το συγκεκριμένο μέσο. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ταμεία πρέπει να παραμείνουν χωριστά και δεν θα πρέπει να υπάρχει επικάλυψη και σύγχυστη ανάμεσα στα δύο. Όχι λοιπόν συγχρηματοδότηση 75%. Για την παράγραφο 9... Χαίρομαι που ο εισηγητής κάνει την πρόταση να γίνει το ταμείο αυτό διαρθρωτικό μέσο, διαρθρωτικό ταμείο. Ας αφήσουμε όμως μια θύρα ανοιχτή, έτσι ώστε το μέσο αυτό να μπορέσει βασικά να γίνει μόνιμο. Θα δούμε τι θα συζητήσει και η προσωρινή Επιτροπή για τις Δημοσιονομικές. Έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας πριν πάρουμε κάποιες τελικές αποφάσεις. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 24η Ιουνίου. Έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε όλα αυτά πιο προσεκτικά, να πείσουμε τους συναδέλφους που είναι σκεπτικιστές ότι το ταμείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Και όπως είπε και η συνάδελφος από την Κοινωνική Επιτροπή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είναι γνωστό το ταμείο αυτό, να φαίνεται το ταμείο αυτό, γιατί σας διαβεβαιώ ότι στην Ιταλία το ταμείο αυτό είναι άγνωστο και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Αγαπητή Μπάρμπαρα, δεν έχουμε πάντα ανθρώπους που να διαφημίζουν το ταμείο αυτό της δικής σας ποιότητας. για να, πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσει τη συζήτηση, μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, με πολλές συγκλήσεις αλλά και αποκλήσεις και διαφωνίες, να κάνω δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Η εμπειρία αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη για το μέλλον. Ανεξάρτητα από την τελική μας θέση. Γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές παρέμβασης και η διάγνωση η οποία βγαίνει από την ανάλυση της κάθε περίπτωσης μας δείχνουν τις ατέλειες των προηγούμενων θα έλεγα μεθόδων που ακολουθήσαμε. Όπως είπε η κυρία Σαρτιέ, υπήρχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ήταν καταρτισμένοι, δεν ήταν επαρκώς ικανοί να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις. Συνεπώς θα υπάρξουν αρκετά συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε σε σχέση με τα κοινωνικά προγράμματα, με τα μόνιμα διαρθρωτικά προγράμματα από τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Το δεύτερο πράγμα στο οποίο να επιμείνω, τα είπε η Μπάμπαρα Ματέρα, όπως επίσης και η κυρία Τρούπελ. Και ο κύριος Μπόκρος επίσης είπε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά ανακατεύεται με τέτοια θέματα. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ε, έχει θα έλεγα πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα. Στην ουσία δηλαδή συγκεντρώνουμε τα φώτα σε μία μορφή έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείχνουμε ότι όταν έχετε πρόβλημα σας βοηθά το κράτος σας, το κράτος μέλος, αλλά παρόλα αυτά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οικογένεια η οποία εκφράζει την αλληλεγγύη της. Η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι ότι για να εκφραστεί αυτή η μορφή αλληλεγγύης θα πρέπει να εκπληρούνται μία από τις εξής δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχουν χρήματα. Χρήματα εμείς σε αυτή τη φάση δεν έχουμε. Δεύτερη προϋπόθεση, να είμαστε σε θέση να φανούμε γενναιόδοροι με χρήματα άλλων. Αυτό είναι πράγματι μια ικανότητα την οποία έχουν οι Αμερικανοί φίλοι. Παντού όπου βάζει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένας Αμερικάνος επίσημος ο οποίος φτάνει και βάζει από πάνω την Αμερικανική σημαία και όλοι ευχαριστούν τις Ηνωμένε Πολιτείες σε πολλά μέρη. Εμείς λοιπόν σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε σημεοφόρους. Αλλά πού είναι οι σημεοφόροι αυτοί, στις Βρυξέλλες στα γραφεία τους. Λοιπόν, έχει σημασία αυτό. Πρόκειται για ένα πολιτικό πρόγραμμα λοιπόν. Είναι καθαρά πολιτικό με την καλή έννοια του επιθέτου αυτού. Βιώνουμε μια κρίση οικονομική σε μια δύσκολη στιγμή και πρέπει να αποδείξουμε την αίσθηση της αλληλεγγύης της κοινωνικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς χρήματα. Και αν οι χρηματαγορές αμφισβητούν για την οικονομική μας ε, ε, υγεία θα έλεγα και αν ένα κράτος μέλος βιώσει σημαντικές δυσκολίες, είδατε πόσος χρόνος χρειάστηκε για να βρεθεί μια κάποια λύση για το ελληνικό πρόβλημα, αυτό σημαίνει γιατί δεν έχουμε έναν ικανό προϋπολογισμό για να καλύψει τα απρόβλεπτα. Κάθε φορά που δημιουργείται μια πρόκληση πρέπει να αποθήξουμε ότι είμαστε ε, ικανοί να σταθούμε αλληλέγγυα ένα στον άλλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία βέβαια ότι στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Midterm Review η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει να δεκαπλασιαστεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός, αλλά εν τω μεταξύ όμως Εν τω μεταξύ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαδικασίες αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας χρησιμοποιώντας την πολιτική διάσταση ε, γνωρίζοντας και τα οικονομικά εμπόδια. Αυτά λοιπόν. Ίσως να ξεκινήσει η Ελίζαμπετ και μετά να κλείσει ο κύριος Πόρτας. Κύριε Σαρτιέ. Ευχαριστώ. Με μεγάλη ενδιαφέρον άκουσα όλα όσα είχαν να πούνε οι συνάδελφοι. Αλλά θέλω να επανέλθω στο εξή σημείο. Ναι, πρόκειται για πρόγραμμα κάτι επίγον που το χρειαζόμαστε. Χρειάζεται να υπάρξει αυτή η προβολή. Και όπως είπε η κυρία Τρίπελ, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορέσουμε να προχωρήσει η υπόθεση της απασχολησιμότητας των ε, και γι' αυτό δεν θέλουμε βέβαια ταυτόχρονα να εγκαταλείψουμε τις άλλες βασικές μας ε, πολιτικές που εκπηγάζουν από την πολιτική για το 2020, από την πολιτική της Αττικής της Λισαβόνας. Αυτό που θέλουμε είναι να αναβαθμίσουμε την ε, κατάρτιση που παρέχεται ούτω ώστε σε τακταδιαστήματα να καταρτίζονται οι εργαζόμενοι ε, με τρόπο έγκυρο και έτσι να μπορούν να είναι πιο προσαρμοστικοί. Άρα θα πρέπει να δούμε τι άλλο χρειάζεται, τι συνοδευτικές πολιτικές θα πρέπει να βρεθούν για διέξω από την κρίση και τέτοιες πολιτικές να ασκήσουμε. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται πέραν των πολιτικών ουσίας και κάποιες άλλες πολιτικές κατεπηγούσης φύσεως. Αυτό το λέγαμε και αυτό θέλουμε και ολοκληρώσει κατάρτιση. Αυτό χρειάζεται. Τώρα όσον αφορά την εξατομικευμένη δράση βεβαίω και για δύσκολη υπόθεση. για την κατάρτιση, για την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται, γιατί ακριβώς η μαζική, μαζικά σκούμενη πολιτική δεν ωφελεί και γι' αυτό και παράλληλα με τις πολιτικές και τα προγράμματα τα οποία είναι δόκιμα, τα οποία είναι επιμέτρο, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και κάποιος ράφτης του ΣΥΠΗΝ ο οποίος να προσαρμόζει την κατάσταση ή στις δυσκολίες τις συγκυριακές. Όσο αφορά αυτές τις υποψίες που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, εγώ είμαι μέλος για που ε, μελετά όλες εξέλιξεις από το που γεννήθηκε αυτό το ταμείο. Γι' αυτό και θέλω να σας καθησυχάσω ότι αυτή η ομάδα εργασίας δουλεύει εις Και όπως ανέφερε ο πρώτος Λαμασούρ, πρόκειται για πολύ καλά εξοπλισμένη ομάδα. Απλά βάσεων. Και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε από τη μία μεριά για αυτό το ταμείο τι γίνεται με, με τα θέματα που υπάρχουν στην ομάδα εργασία και από την άλλη μεριά όμω να δούμε πέραν των θεμάτων, πέραν τη θεωρία, να δούμε στην πράξη τι γίνεται και έτσι να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Οπότε και στην Επιτροπή Γενικών Υποθέσεων ε, με αυτό το πνεύμα συντάξαμε και υποβάλλουμε κάποιες τροπολογίες για να δούμε πώς βέβαια θα καταλήξουμε σε συνδυασμό και έτσι να υπάρχει ομοιογενής ε, οπτική για το μέλλον αυτού του ταμείου και όλα αυτά να συντεριάξουν στο γίνεται καλύτερα με το σώμα της εκθέσεως του κυρίου Πόρτας. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε κύριε συνάδελφε. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια της ε, Κοινωνικής Επιτροπής, την κυρία Μωρόν Σορτιέ, για τη βοήθεια που μου παρέσχει, αλλά να ευχαριστήσω και όλη την Επιτροπή Απασχόλησης. Εγώ εξήγαγα τα, ό,τι σήμερα εξήγαγα επί τη βάση του υλικού που μου παρέσχε η ομάδα εργασία αυτή. Βέβαια, με απασχόλησαν πάρα πολύ και τα δημοσιονομικά ζητήματα. Μια που κυρίως αρμόδια είναι η δική μας επιτροπή. Την πρώτη φορά που έλαβε το λόγο ο κ. Λαμασούρη είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι θα πρέπει να δούμε Μήπω και το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να καλύψει τα θέματα που καλύπτει τα θέματα του Ταμείου της Παγκοσμιοποίησης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα γιατί τώρα αυτό το οποίο συζητούμε είναι το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα υπόλοιπα. Ταμεία. Και τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος. Γιατί υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες, κάποιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και έχουμε ένα σωρό ταμεία και δεν μπορούμε όλα μαζί να τα στριμώξουμε σε μία και μόνη συζήτηση όπως αυτή που κάνουμε σήμερα για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό σε απάντησα αυτό που είπε ο πρόεδρος. Έχω να πω ότι βρισκόμαστε στην κλασική περίπτωση που το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Αν δηλαδή το Ταμείο Προσαρμογής στη Μεξονοποίηση το διασπάσουμε και κοιτάξουμε τα 27 χωριστά προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου, δεν θα βγάλουμε τίποτα. Δεν θα έχουμε εγγυήσει για το ότι θα βοηθηθούν καλύτερα οι απολυθέντες με τις ομαδικές απολύτες. Ότι θα έχουν καλύτερη μεταχείριση από τα εθνικά προγράμματα, τα 27, σε σχέση με αυτά που τους καλύπτει τώρα το Ταμείο της Παγκοσμιοποίηση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν εγγύσεις ποιότητα σε αυτό το ταμείο. Ούτως ώστε να μπορεί κανείς να ξανενταχθεί στον επαγγελματικό του κλάδο. Καλά, δεν αφορά αυτό όλους τους ανέργους, αλλά κάποιους. Αυτούς που έπεσαν θύματα ομαδικών απολύσεων από μεγάλες εταιρείε ή σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. αυτή τον οποίων υπέστη πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα η ζωή λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όπως είπε και η κυρία Τρίπελ θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε όπως γίνεται κάθε φορά που συζητάμε το αν θα πρέπει να σταματήσει ένα ταμείο. Θα πρέπει να κάνουμε έναν ισολογισμό αν είναι αρνητικός ή θετικός. Και σε αυτή την περίπτωση είναι αρνητικός. Είναι κακό να σταματήσει να υπάρχει αυτό το ταμείο. Να, και άλλη μια διαφορά μεταξύ του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και του Κοινωνικού Ταμείου. Για τις υποψηφιότητες εν προκειμένου μπορεί να ασκήσει πολύ καλύτερο πρόγραμμα, η, πολύ καλύτερο έλεγχο η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά στα πολιετή προγράμματα των κρατών μελών. Η διασπάθηση επομένω του κοινοτικού χρήματος, κατά τη γνώμη μου, φρενάρεται πολύ περισσότερο στα πλαίσια του αυτού παρά στα 27 προγράμματα του κοινωνικού ταμείου. Άρα, εδώ δεν έχουμε χρήματα τα οποία διασπαθίζονται και πάνε χαμένα. Δεν λέμε για χρήματα από τον προπολογισμό. Μιλάμε για κάποιους πόρους που είναι εκτός προπολογισμού. Χρήματα που αξιοποιούνται και ξανααξιοποιούνται όταν δεν απορροφούνται στην προηγούμενη χρήση. Γι' αυτό δεν χάνονται χρήματα παρά μόνο εάν δεν έχουμε την επιστροφή διότι κάτι διέφυγε του ελέγχου των αρμοδίων αρχών. Κάτι άλλο σημαντικό. Αυτό που είπε ο κύριος Γκαρίγα σε σχέση με την επικουρικότητα. Μεταξύ δηλαδή δράσης Ένωσης και κρατών μελών όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές. Είναι ένα επαρκτό πρόβλημα. Όμως δεν μιλούμε εδώ για ένα υποχρεωτικό ταμείο. Μιλάμε για ένα ταμείο συμπληρωματικό όσον αφορά την κυρίαρχη ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών για κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόληση. Δεν είναι υποχρεωτικό παρεμβαίνει μόνο όταν το ζητήσει κάποιο κράτος μέλος, γιατί το θέλει το κράτος μέλος για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση κατάσταση. Ούτε μπορεί, ούτε, ούτε πρέπει να έχει διαρκή χαρακτήρα γιατί ακριβώς αφορά εξαιρετικές περιστάσεις. Τέλος αυτό δεν ισχύει απόλυτα. αυτό το ταμείο κινητοποιείται σε συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Ξέρετε, δεν κλείνουμε ραντεβού ούτε με το τσουνάμι ούτε με τον ε, σεισμό. Άρα αντίστοιχα και για το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το έχουμε, ούτω ώστε να έχουμε χρήματα αν συμβεί το εξαιρετικό, το τσουνάμι ας πούμε. Αυτό ισχύει και για τις ε, συλλογικές, ομαδικές απολύσεις. Πρόκειται για κάτι το οποίο πλήσει πολύ πολύ το κοινωνικό ιστό αυτέ οι ομαδικέ απολύσει. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο επίση σοβεί ακόμα και σε περίπτωση ανάκαμψη της οικονομίας. Άρα, να, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο ταμείο και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Γιατί είναι φαινόμενοι απολύσεις διαρκές δυστυχώς. Η Χέλγα πάρα πολύ σωστά είπε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, θα μπορούσαμε να έχουμε αντί αυτό το ταμείο, βελτίωση των υπαρχών των ταμείων. Υπάρχουν κάποιοι εδώ που είναι πάρα πολύ παλιοί. Εγώ είμαι φρέσκο σχετικά και ξέρετε καλύτερα εσεί ε, τόσα χρόνια πώ καταρτίζεται ο προπολογισμό. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν δυσκολίε συντονισμού μεταξύ των επιμέρου προγραμμάτων όταν έρθει η ώρα τη εκτέλεση επιτόπου. Θα πρέπει να επιληθούν αυτέ οι δυσκολίε, Αλλά δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε για κάθε περιφέρεια, κάθε περιοχή άλλο πρόγραμμα. Έχουμε ένα σωρό προγράμματα. Και με αυτό το ταμείο για τη Μεγισμιοποίηση θα μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα του να έχει την ισόβια κατάρτιση. Άλλο πρόβλημα αυτό. Αυτό κάνω εγώ. Θέλω να υπάρχει κάτι που να καλύπτει του εργαζόμενου σε κάτι που πολύ, πολύ συγκεκριμένε καταστάσει, οι οποίε δυστυχώ είναι πάγιε. Συμβαίνουν συνεχεί, συνεχώ, όπω αυτέ οι σημαντικέ απολύσει. Νομίζω ήταν πάρα πολύ πλούσια αυτή η συζήτηση. Και πάρα πολύ ωραία τα είπε ο κύριο Νταρντέν. Όπως τα είπε για, για, την, ε, για, για, το γιατρό, τον οικογενειακό γιατρό από τη μία και την άλλη μεριά τα κατεπήγοντα των νοσοκομείων. Αυτή ήταν πολύ ωραία εικόνα. Χρειάζεται λοιπόν και ο γιατρός και το νοσοκομείο τα κατεπήγοντα. Βέβαια, το 2013 θα, θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα μπορούμε συνέχεια να ε, κάνουμε το ίδιο την πρικοδότηση αυτού του ελέγχου, αυτού του ταμείου. Και ε, θα δυσκολεύει ο Λένα ο έλεγχος του προπολογισμού. Αλλά το κόστος των επολύσεων θα ε, είναι τέτοιο από το οποίο θα εξαρτάται η πρικοδότηση του Ταμείου. Όπως είναι τώρα η κατάσταση, κανείς δεν ωφελείται. Βαρύνεται ο προπολογισμό και όπως είπε ο κ. Λαμασούρ, πρόκειται για δημιουργική τεχνική που τώρα χρησιμοποιεί. Σας ευχαριστώ τον συγητή και όλους τους Θα ε, Ήταν πάρα πολύ εμπλουτιστική αυτή η ανταλλαγή απόψε σας. Υπενθυμίζω η για την αποβολή των απολογιών 24 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Την ίδια μέρα η Επιτροπή Απασχόληση θα υιοθετήσει τη δική της γνωμοδότηση και στις 13 και 14 Ιουλίου θα εγκρίνουμε την σχέδιο έκθεση ενδεχομένω μετά από προετοιμασία συμβαστικών τροπολογιών. Στην Ολομέλεια θα περάσει το θέμα αυτό για ψηφοφορία στην πρώτη σύνοδο του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, χρονοτρυφήσαμε κάπως, άξιζε το κόπο μας, θα επιταχύνουμε λίγο, θα παραμείνουμε στο προβλησμό 2011 με τον σημείο 10. Ο κύριος Ιβαϊλό Κάλφιν θα μας δώσει την αποψή του για χωρίς εγγύηση της Ευρωπαϊκής στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη μειών από δάνεια και εγγύηση για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρο, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να κάνουμε κάτι που ακολουθεί μία απόφαση της ε, Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας ε, για την χωρίς εγγύησης για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας της Κοτονού. Οι συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε συμπεριλάβονται σε έγγραφα που έβαλε η Κομισιόν, πρόκειται για έκθεση της Κομισιόν και θα ε, θέλατε ίσως να δώσετε το, λόγο μετά στον κύριο Καζάνη, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν εδώ κύριε Πρόεδρε, για να μας διαφωτίσει καλύτερα όσον αφορά αυτά τα κείμενα. Κατά βάση, Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά προσδημασία των εγγράφων αυτών η Κομισιόν χρησιμοποίησε δύο διαδικασίες θα έλεγα για να προετοιμάσει το, το έγγραφο. Υπήρχε μια ομάδα σοφών στους οποίους πρόεδρε ο κ. Μισελ Καντεσιού Και η ομάδα αυτή έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα εις βάθος αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που οπωσδήποτε θα συζητηθούν εις βάθος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαι σίγουρος. Και υπήρχε ένα κείμενο το οποίο παρουσίασαν εξωτερικοί σύμβουλοι. Ποια είναι τα προβλήματα που εξευρέθησαν στις ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην περιοχή αυτή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέχρι σήμερα. Καταρχήν, υπήρχαν πολλές διαφορές μεταξύ των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μια που η τράπεζα αυτή είναι μια τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καμιά φορά είχαμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιούσε πλήρως όλα τα μέσα που είχε για τα μέσα αυτά. Η δεύτερη κριτική που παρουσιάζεται είναι όταν εκπρόσωποι μη κυβερνητικών των οργανώσεων Ε, βρέθηκαν στο προσκήνιο και πρόκειτο για τους ε, στόχους των ανάπτυξης. Ε, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργήθηκε για να κάνει επενδύσεις. Γι' αυτό οι προσδοκίες που υπήρχαν μέχρι στιγμής ήταν υπερβολικές. Αυτή είναι μία από τις κυρίες ανησυχίες ε, της κοινότητας και των διαφόρων ε, εμπλεκομένων, οπωσδήποτε. Επίσης, υπήρχε το θέμα της χρήσης διαφορετικών μέσων σε διαφορετικές περιφέρειες. Δεν υπήρχε δηλαδή συνέπεια όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στι διάφορες περιφέρειες. Μετά υπήρχε το θέμα για την πρόσβαση στους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καταρχήν ξεκίνησε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόθεση των ευρωπαϊκών επενδύσεων εκεί. Αργότερα ασχολήθηκε με θέματα ανάπτυξης ό,τι φορά λοιπόν η χρήση πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν ανταποκρίνεται στι ανησυχίε για την ανάπτυξη. Παρόλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα ρόλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι να ενθαρρύνει τι επενδύσει από ευρωπαϊκέ τράπεζε στι περιφέρειε αυτέ εκτό Ευρώπη. Πάντα βέβαια υπάρχει το πρόβλημα της ισορροπίας μεταξύ των καθαρά τραπεζικών δραστηριοτήτων και του πολιτικού ε, συμφέροντος. Και εδώ οφείλονται ορισμένες από τις διαφορές. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μία τράπεζα. Και πρέπει να ακολουθεί τις διατάξει που διαπούν αυτού του είδου του ε, οργανισμούς. Και τέλος, Θα ήθελα να σας πω ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα του τελευταίου μήνε. Είναι η συνεργασία με τι Ευρωπαϊκές Τράπεζες Επενδύσεων και των Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών, παραδείγματο χάρη συνεργασία με την Διεθνή Τράπεζα, ε, ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανάπτυξη, τη δυνατότητα συνεργασίας ε, βασιζόμενη σε δωρεές της Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να είναι εξαιρετικός αυτός είναι ο κατάλογος των κύριων θεμάτων των τελευταίων μηνών, όπου έλεγε χώρα η προετοιμασία αυτή τη ε, μεσοπρόθεσμη ε, αναθεωρήση. Τώρα έχουμε μπροστά μα την πρόταση τη Κομισιόν. Σε μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα, καλύπτει πολλέ από τι ανησυχίε μα. Η πρόταση Κομισιόν είναι να Παραταθεί η εντολή μέχρι το 2013 και να συμπεριληφθούν νέα στοιχεία, ούτω ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναποκρίνεται καλύτερα στι προσδοκίε που υπάρχουν. Αυτό προτείνεται, όπως σας είπα, να παραταθεί η εντολή μέχρι το 2013, να δοθούν 2 δισεκατομμύρια ε, ευρώ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο υποθεματικό και αυτά δύο δις να κατακτηθούν σαν ένα μέσο για την ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα των ε, κλιματικών αλλαγών. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν μόνο τροπαθήσεις όσον αφορά τις δέσεις στον τομέα των κλιματικών αναλογών. Ίσως αυτά τα δύο δις θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Η πρόταση επίση έχει μια σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κοινωτικών πολιτικών και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. ε, προσπαθώντας έτσι να επιτευχθεί και μεγαλύτερη ευελιξία σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν ε, πολλές νέες χώρες που συμπεριλαμβάνονται Και υπάρχουν και πολλές προτάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να δράσαν ένα ε, μέσο της πρόθεσης της πολιτικής ανάπτυξης. Ναι. Μπορούμε να δούμε κατά πόσον οι στόχοι που αναφέρει η Κομισιόν είναι αρκετά φιλόδοξοι, κατά πόσον ε, τα προβλήματα θα ληφθούν με το 2013 ή κατά πόσο θα πρέπει να δούμε πώς θα αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις περιφέρειες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Ε, πρόκειται για θέματα που το θα συζητηθούν ε, έντονα. Να συγκεντρωθούμε περισσότερο στους στόχους ανάπτυξης. Αυτή είναι η κύρια ανησυχία των συναδέλφων μας στην Επιτροπή Ανάπτυξης που έχει κάνει μια αναλυτική ε, εξέταση της, του έργου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο κ. Καμπτεσί προτείνει να υπάρχει μια νέα τράπεζα για τα θέματα της ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτό το 2013, όσο μπορούσαμε κάτι να προετοιμάσουμε. Αυτό είπε, είναι θέμα που θα πρέπει να ελέγξουμε εις βάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κόστος μιας τέτοιας ε, εξέλιξης. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται στην έκθεση Καμπτεσίου και θα είναι ένα θέμα υψηλού ε, ενδιαφέροντος στο Κοινοβούλιο. Ο λεγόμενος μηχανισμός ένταξης, blending mechanism, που θα μπορέσει οπωσδήποτε να βοηθήσει. Υπάρχουν πολύ καλές εμπειρίες, πολύ καλά παραδείγματα για την εργασία της τράπεζας σε ορισμένες περιφέρειες, αλλά πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν για να δημιουργηθεί ο σωστός μηχανισμός που θα δημιουργήσει τις συνέργειες αυτές. Μετά είναι το θέμα της εργασίας με τους άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Προτείνεται να δημιουργηθούν κάποιες πλατφόρμες όπως λέμε. Είναι καλή ιδέα, αλλά όταν φτάσουμε στις λεπτομέρειες βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και θα πρέπει να δούμε τις μέχρι τότε εμπειρίες ε, να τις αναλύσουμε για να δούμε πώς θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Τέλος, συνδεσμός με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να είναι νομίζω ένα από τα κύρια θέματα στην ε, αναθεώρηση αυτή που κάνουμε σήμερα. Γιατί από τα στιγμικά στοιχεία βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι πολύ και σε ορισμένε περιφέρειε, στι χώρε τη προομεθρικέ, στην Ανατολική Ασία, όχι όσον αφορά του ανατολικού μα ε, εταίρου, ε, την Ρωσία Φερρυπίν. Και όταν εξτάζουμε του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι διάφορε περιφέρειε αυτέ, ενδεχόμενη σύγκληση των ε, οικονομιών, παραδείγματο χάρη στι προενταξιακέ χώρε, κλιματικές αλλαγές όπως είπαμε παντού κλπ. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τέλος, για να ολοκληρώσω αυτές τις αρχικές έτσι κάπως αφήσει ιδέες, προτείνουμε ένα χρονοδιάγραμμα που το έχετε μπροστά σας, στο Combo News η ιδέα είναι να θεωρήσουμε τη γνωμοδότηση αυτή το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή να ζητήσουμε τις γνωμοτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων ε, επιτροπών τον Οκτώβριο με τη σκέψη να προσπαθήσουμε να ε, εγκριθεί η έκθεση στην Ολομέλεια πριν από το τέλη του έτους. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Συμβούλιο, υπάρχει διαδικασία δεύτερης ε, διαλλαγής αρχές του επόμενου έτους αλλά αν δεν το εθετήσουμε μέχρι τα μέση του επόμενου έτους ε, το έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στις περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να καθυστερήσουμε υπερβολικά και να περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Το πρόγραμμα που προτείνεται έχει σαν στόχο να καταστήσει τα πράγματα δυνατά για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η έρευξή μας μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε, ευχαριστώ για μια ξεκάθαρη αλλά και συνθετική παρουσίαση. Je vous propose de ne pas... Θα ήθελα να σας προτείνω να μην συζητήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό σήμερα. Έχουμε ένα πρόβλημα τώρα στην ημερήσια διάταξη. Έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεως, απόψεων κατά την παρουσίαση του κυρίου Καμτεσού. Είχε έρθει ε, πριν λίγους μήνες να παρουσιάσει και ήταν πρεμιέρα θα έλεγα γιατί δεν το είχε παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα. Όπως είπε ο εισηγητής μας ε, και άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδιαφέρονται. Δύο από αυτές, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Ανάπτυξης, θα ήθελα να συνεργαστούν μαζί μας επί τη βάση του άρθρου 50, 51, 52, 53 και ούτω καθεξής. Η λύση την οποία προκρίνουμε σε συνεργασία με τον εισηγητή είναι όπως και να έχουν τα πράγματα. Εμείς παραμένουμε η Επιτροπή επί της ουσίας. Οι εισηγητές για γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης συμμετέχουν και θα υπάρξουν κοινέ προτάσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο μας παρουσιάστηκε πριν από λίγο. Δηλαδή το Σεπτέμβριο να εξετάσουμε μία πρώτη γραπτή έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ενώ οι άλλες επιτροπές θα ασχολούνται με τις νομοδοτήσεις τους, να υιοθετηθεί η έκθεσή μας στις 9 Νοεμβρίου και αν πάνε όλα καλά να ψηφίσουμε το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια. Όλοι θέλουμε να υπάρξει μια απόφαση πριν το τέλος του χρόνου γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει προετοιμαστεί σωστά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερήσει κανείς ε, επί μακρόν το θέμα. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Καλφίν. Σας ζητώ να περάσουμε ταχύτατα στον προϋπολογισμό του 2010. Έχουμε πολλά σημεία τα οποία θα εξετάσουμε συνοπτικά. Το σημείο 11, διορθωτική επιστολή παρίθμου 2 ο εισηγητή μα δεν είναι εκεί, αλλά ούτε και το θέμα, οπότε μπορούμε να τελειώσουμε γρήγορα. Πρόκειται για τα συμπληρωματικά μέσα, τα οποία ζητήθηκαν από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική για να καλύψουν τι νέε αρμοδιότητε τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει σχετικά με τα θέματα αυτά. Εφόσον δεν προχωρά το Συμβούλιο λοιπόν, ούτε και εμείς μπορούμε να πάμε πουθενά. Περνάμε λοιπόν άμεσα στο σημείο 12 είναι το θέμα της μπανάνας ουσιαστικά. Πώς έχουν γενικά οι συζητήσεις γύρω από το θέμα της μπανάνας κύριε Σούριανα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμένα η θέση μου παραμένει η ίδια με το παρελθόν. Από ό,τι γνωρίζω θα υπάρξει τριμερής διάλογος για το θέμα αυτό θα δούμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ή όχι μια κάποια θέση. Η πρώτη αντίδραση του Συμβουλίου ήταν ε, μηδέν. Τίποτα από το μέσο ευελιξίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μετριοπαθής και αρκετά χαμηλή σχετικά με το ποσοστό του μέσου. Μιλάμε ότι το θέμα αυτό είναι χαρακτηριστικό θα έλεγα των περιπτώσεων αυτών. Δεν ήταν στον αρχικό προϋπολογισμό του 2010. Οπότε τίθεται το θέμα εδώ της ευελιξίας. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να εμείνουμε στο μηδέν του Συμβουλίου πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από εμά που είναι το 100% και θα ακολουθήσει η διαδικασία συνδιαλλαγής. Θα δούμε τι προτάσεις θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ είμαι έτοιμος να, να εφαρμοστεί όχι το μέσο ευελιξίας, ενώ να είμαι πιο ευέλικτος. Είναι διοντολογικά απαραίτητο να προχωρήσουμε Έχουμε ευθύνες απέναντι σε χώρες που έχουν πολύ σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα. Ιδιαίτερα επειδή εμείς οι ίδιοι παράγουμε ένα ποσοστό αυτών των δυσκολιών. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση όχι απλά να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, αλλά να υπάρξει ε, μια κάποια πειθαρχία σε σχέση με τα δημοσιονομικά πριν οποιοδήποτε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο όνομα της Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις και δώσει υποσχέσει χωρίς συγκεκριμένη εντολή από τις αρχές επί του προϋπολογισμού. Κατανοώ τη θέση λοιπόν του Συμβουλίου, αλλά είναι αδύνατο όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν ενάντια στα συμφέροντα και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δεν είναι δίκαιο, δεν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές της αρχής επί των δημοσιονομικών. Και αν τυχόν είμαστε έτοιμοι, τότε θα είμαστε υπερήφανοι που θα σταθούμε γενναιόδωρα απέναντι στους παραγωγούς πανάνας, αλλά αν η συμπεριφορά αυτή μετατραπεί σε μια συνεχή πρακτική, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο θα παραμείνει απλά ένα τμήμα της αρχής επί του, επί του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα γοήτρου, είναι θέμα του να γίνουν τα πράγματα σωστά. Ελπίζω η συνδιαλλαγή να καταλήξει, να είναι καρποφόρα, αποδοτική και περιμένουμε καινούργιες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω η θέση της Επιτροπής να κατατεθεί κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου και θα δούμε τι δυνατότητες διαχείρισης του θέματος θα έχουμε τότε. Λοιπόν, δεν θα γίνει συζήτηση σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει λόγος να γίνει συζήτηση σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ κύριε Σούριαν. Ο Χάιμε θέλει κάτι να προσθέσει, όχι. Το πολιτικό θέμα. Νομίζω ότι ήδη είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό θέμα. Το πολιτικό θέμα το έχουμε μπροστά μας θα έλεγα. Είμαστε έτοιμοι λόγω αυτής της τεράστιας διαφοράς ανάμεσα σε μας και το Συμβούλιο. Είμαστε έτοιμοι έλεγα να καταστήσουμε το θέμα αυτό θέμα σύγκρουσης και στην ουσία να πάρουμε τις χώρες που τις απασχολεί το θέμα να τις κάνουμε ομήρους θα έλεγα. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε αρνητικά. Αναγνωρίζουμε ότι απέναντι στις χώρες αυτές ε, είναι πολιτικά ανέφικτο το να καθυστερήσει κανείς και το να κερδίσει απλά κάποιος λίγο χρόνο δεν θα βοηθήσει κανένα ούτε τις εμπλεκόμενες χώρες ούτε εμάς. Ο μηχανισμός βοήθειας είναι τέτοιος που ακόμα και αν κάποια στιγμή δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα καλή κατάσταση στο εμπόριο της μπανάνας, δεν θα λυθεί το πρόβλημά μας, θα παραμείνει η εκκρεμότητα. Γιατί αυτό θα αντισταθμίσει το ότι οι συγκεκριμένες χώρες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΠΟΕ, έχουν δικαίωμα, θα έλεγα, σε μια δημοσιονομική αύξηση γιατί δεν χαίρουν των εμπορικών πλεονεκτημάτων τα οποία είχαν στη διάθεσή τους στο παρελθόν. Λοιπόν, επόμενη φάση ο τριμερής διάλογος. Είτε από τον τριμερή διάλογο είτε από ενδιάμεσες διαπραγματεύσεις θα υπάρξει μια θέση συνενετική ανάμεσα στις δύο ακραίες θέσεις τις οποίες σε αυτή τη φάση εκφράζει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτά. Λοιπόν, κλείσαμε και με το 13. Για τον προϋπολογισμό του 2010 θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Καλφίν να μας μιλήσει για μία τροπολογία σχετικά με τον κανονισμό του 2006 για τις... Α, για τις μπανάνες είναι και το 14, sorry, για τις μπανάνες και το 14, οπότε δεν θα μας πείτε κάτι για τις μπανάνες. Λοιπόν, την μπανάνα τη φάγαμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η ούτε θα πάρει το λόγο για τον οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων συστημάτων πληροφορικής. Ιούτα. Ευχαριστώ. Είδες η περισμένη μας συνειδρίαση συζητήσαμε το θέμα για μακρόν Είχα υποβάλει κάποιες ερωτήσεις προς την Κομισιόν, απαντήθησαν ανεπαρκώς. Εν τω μεταξύ όμως είχα διάφορες ε, συναντήσεις με τους αρμοδίους της Κομισιόν και με συνεργάφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και η πρότασή μου υπάρχει τώρα για μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων. Εμείς ε, πρέπει να περιορίσουμε την προσοχή μας στην υποβολή τροπολογιών οι οποίες υπάρχονται βέβαια στις δικές μας αρμοδιότητες. Και αυτό παρόλο υπάρχουν πολλές τροπολογίες, εγώ υποβάλλω 24, περιορίστηκα όμως πραγματικά μόνο στις δημοσιονομικές πτυχές της υπηρεσίας αυτής πληροφορικής. Και πρέπει να πω ότι δεν έκανα εγώ ε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ο εισηγητής εκεί στη γνωμοδότηση επικρίνει γενικά και την νομική βάση της εν λόγω υπηρεσίας κλπ. Δεν είναι αυτό νομίζω αρμοδιότητά μας. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι σε ορισμένα σημεία θέλουμε να αλλάξουμε ουσιαστικά αυτή την ε, ε, υπηρεσία στην περίπτωση κατά οποία θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους της ε, Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Στάνφος Κοέλιο στην Ελλόγου Επιτροπή είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος και αν κάποιος από εμάς έχει καταπληκτικές ιδέες, είμαι σίγουρη ότι θα τις, ε, θα τις συμπεριλάβουμε. Αλλιώς θα πρέπει εμείς να περιοριστούμε στις επιφυλάξεις που έχουμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών. Οι δικές μου 24 τροπολογίες έχετε απαριθμίσει στη σελίδα 5 και λέμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι χρειάζεται. Ελέγχθη ό,τι έπρεπε να δεχθεί για την υπηρεσία αυτή. Παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα που είναι γενικά και όπου οπωσδήποτε δεν θα επιληθούν τώρα από την Κομισιόν. Πρώτα για τα θέματα που έχουμε πάντα να θίξουμε όταν από τους λειτουργικούς πόρους ε, χρηματοδοτούμε διοικητικές εργασίες. Ακριβώς αυτό γίνεται και εδώ. Ξέρουμε, όπως το προτείνει και η Κομισιόν, πώς εντάσσεται αυτό στον προγραμματισμό χωρίς να ξεπερνάει τα όρια του προπολογισμού μας γιατί υπάρχουν χρήματα από άλλα κονδύλια τα οποία μεταφέρονται εδώ. Μάλλον λοιπόν δημοσιονομικά δεν υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον όχι μέχρι το 2013. και αν συμφωνήσει η Επιτροπή Εσωτερικών για τη δημιουργία αυτού του τύπου της υπηρεσίας δεν είναι 100% σίγουρο, αλλά αν συμφωνήσει μπορούμε εμείς με τη δική μας γνωμοδότηση να συμβάλλουμε τους ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι δημοσιονομικές πτυχές και να ενταχθούν επίσης στα εν λόγω κείμενα. Στα Κόμπου νιούς ε, αναφέρεται ακριβώς ε, και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τι είναι, α, 24 Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι. 13 Ιουλίου θέλουμε να ψηφίσουμε και θεωρούμε ότι το Σεπτέμβριο η Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων θα εντάξει τη δική μας γνωμοδότηση στη δική της έκθεση. Γιούτα, σε ευχαριστώ. Αλλά ο κύριος Κολίνο έχει δει στο λόγο. Σαν σκιώδη στη για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα ήθελα να υπογραμμίσω την θετική δουλειά της εισηγήτριας και να εκφράσω και κάποιες σκέψεις. Η υπηρεσία αυτή θα διαχειριστεί το σύστημα του Σέγγεν και το Eurodac. Βασικός στόχος λοιπόν της λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής είναι να διαχειριστεί σωστά αυτούς τους τομείς και να διασφαλίζει την παραγωγή δεδομένων σε 24 ώρη βάση. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας ότι στόχος της υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των στοιχείων η ευθύνη για την επιλογή των στοιχείων είναι θέμα των κρατών μελών, μονομένα κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να συντονίσει τα τρία διαθέσιμα συστήματα η υπηρεσία αυτή, να κάνει οικονομίες κλίμακας, να δημιουργεί ακριβώς τους τρόπους με τους οποίους θα εκμεταλλευόμεθα ε, στο μέγιστο τα διαθέσιμα μέσα με τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει να λειτουργεί ουσιαστικά από το 2012, θα συσταθεί το 2011, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά το σύστημα, το περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013. Τα 113 εκατομμύρια που είναι απαράτητα για τη λειτουργία έχουν ήδη προβλεφθεί από φέτος μέχρι και το 2013 και είναι συμβατά με τις ε, προγραμματικές μας προβλέψεις. Η θέση μας λοιπόν δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τη θέση της εισηγητρίας, της κυρίας Χάουγ. Έχει παρουσιάσει αρκετές λεπτομέρειες η κυρία Χάουγκ, γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή μας δεν καλείται να συζητήσει την καταλληλότητα της απόφασης για την δημιουργία της υπηρεσίας αυτής, δεν μπορούμε παρόλα αυτά να παρά να υπογραμμίσουμε ότι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τεκμηρίωση των επιλογών που οδηγούν στην δημιουργία νέων υπηρεσιών δεν είναι ιδιαίτερα τεκμηριωμένη γιατί ξέρουμε ότι θα μπορούσαν και οι άλλες εξωτερικές υπηρεσίες να κάνουν κάτι τέτοιο ή οι ίδιες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το κάνουν. Αλλά πέρα λοιπόν από τις πιθανότητες ε, θα έλεγα μείωσης ε, των εξόδων για τον έλεγχο και τη λειτουργία των τριών συστημάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να συμπεριλάβει πιο συγκεκριμένα στοιχεία στο εσωτερικό της πρότασής της γύρω από την ανάλυση κόστους ωφέλους των στρατηγικών επιλογών που αφορούν την υπηρεσία αυτή και την επιλογή της έδρας. Σχετικά με την έδρα της υπηρεσίας θα πρέπει να πούμε ότι η επιλογή δεν θα πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά σε παραμέτρους ελκυστικότητας μιας πόλης και να αφήσουμε εκ των υστέρων το κατά πόσον το συγκεκριμένο κράτος μπορεί να καταστήσει την πόλη τη συγκεκριμένη συμβατή με τις ανάγκες και τις απαιτήσει. Απαιτείται να γίνει λοιπόν μια αναλυτική εξέταση όλων των δυνατοτήτων και των εναλλακτικών προτάσεων που υπάρχουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μου άρεσε η αποστροφή της ομιλίας του προλαλήσαντος γιατί θα ήταν πάρα πορεία να μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτό. Στο να μπορούμε έτσι να κάνουμε την επιλογή μας. Φυσικά και το Συμβούλιο κάνει ό,τι θέλει γιατί είναι δική του δουλειά το να αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οργανισμό αυτό να μπορεί να βρεθεί η πόλη που θα κατασταθεί να έχει τις, ε, την υποδομή τι ε, διευκολύνσεις αυτό που είπε η Γιούτα που αντικατοπτρίζουν αυτά που εμείς πάντοτε υποστηρίζαμε τέλος πάντων μου αρέσουν πάρα πολύ τροπολογίες της Γιούτα και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον προπολογισμό μόνο και να μην αρχίσουν να επισέρχονται σε θέματα πέραν του προπολογισμού. Και ο Σάλβαρο, Άλβαρο που σήμερα δεν είναι μαζί μας, επίσης ενδιαφέρεται πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ε, συμμετέχει και αυτό στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Τον ενδιαφέρει πολύ το πώς θα βρεθεί ε, το κράτος που θα υποδεχθεί και θα αναδεχθεί τον οργανισμό και να δούμε πού θα επιφυλαχθούμε τόσο δεν είναι του παρόντος. Καταρχήν πάντως εγώ είμαι υπέρ των 24 τροπολογιών της Γιούτα. Très bien, merci. Ε, Λάμασουρ, πολύ ωραία. Γιούτα, έχεις κάτι να απαντήσεις. Ναι, πολύ σύντομα. Ιδίω πάνω σε αυτά που ελεξαν για την χώρα που θα φιλοξενήσει την προσία. Καλώς Κοέλιο. Στην πρόταση της έκθεσης σου αναφέρει ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει με καμία εξωτερική υπηρεσία εάν δεν αναφέρεται πού πρόκειται να έχει την έδρα της και ότι πρόκειται πραγματικά για την καλύτερη δυνατή έδρα αφού ο σκοπιά εσωτερική πολιτική ίσω είναι διαφορετικό, αλλά αποτελεσματική, πραγματικά καλή έδρα είναι κάτι που μα ενδιαφέρει και εμά. Και είναι αυτό που θέλουμε και εμείς. Ακριβώς όπως όπου αναφέρεται εδώ στο σχέδιο έχει εγγραφεί στην έκθεση. Πρώτη φορά η, ε, ο χρηματοδοτικός προγραμματισμός της ε, Κομισιόν είναι τόσο ακριβής. Θα δούμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Λοιπόν, για τις εργασίες στην έκθεση μας είπε η της η Γιούτα προηγουμένως. Θα έλεγα να ολοκληρώσουμε τώρα την σημερινή μας εργασία με τα σημεία 5, 6 και 7, δηλαδή τις πολιτικές ε, συνέπειες των ε, προφορικών ερωτήσεων που υποβάλαμε στην Κομισιόν για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προβλέψεων και ίσως στα σύντομα μετά να παρουσιάσετε το σχέδιο προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου για τεχνικούς λόγους πάνω στους ίδιους πόρους. Ο Ράιμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Γιατί εγώ διαφορετικά από την συνάδελφο ε, Ιούτα Χάουκ με την γνωμοδότηση έτσι για τι υπηρεσίε. Εγώ θα έλεγα ότι άσχετα από τις προβλεπόμενες τροπολογίες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει ε, με υπηρεσίες να καλυφθούν εκείνες χώρες που μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία υπηρεσία δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το κριτήριο τελικό που έχει ορίσει και η συγγήτρια του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, την περασμένη Τρίτη είχαμε υποβάλει μια προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο, όπως είχε συμφωνηθεί. Στην αρχή της για την προετοιμασία μιας προσωρινής έκθεσης βάσει του άρθρου 180 καθώ 3 του ιστορικού κανονισμού όσοι συνάδελφοι ήταν παρόντες θυμώνται ότι η, ε, ε ήταν παρόν ο Γενικός Γραμματέας του που υπεύθυνος για τον Ισπανικό προπολογισμό, μέρος της ε, Ισπανική Προεδρία. Σήμερα εξέτασα το επιλέξει πρακτικά τη συζήτηση για άλλη μια φορά Και είδαμε ότι βέβαια η Προεδρία του Συμβουλίου βρισκόταν ενώπιον μιας μη ομόφωνης άποψης στο ίδιο το Συμβούλιο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η τελευταία αναλύση χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικά. Ε, θα πρέπει να εξτάσουμε αυτά που είπε ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι. Από τη μια μεριά είπε ξεκάθαρα ότι η Κομισιόν μπορεί να προτείνει μόνο μια αναθεώρηση εάν αυτό είναι πραγματικά αναγκαίο. Κατά δεύτερον όμως είπε ξεκάθαρα ότι τα απαραίτητα μέσα για την ευελιξία, τα περιθώρια και τα αποθεματικά είναι θέματα στα οποία αποκλίνει η Κομισιόν από την άποψη του Συμβουλίου. Είπε μάλιστα ξεκάθαρα ότι όσον αφορά για το άρθρο 8.3 εμείς θέλουμε να προασπίσουμε την ευελιξία αυτά είναι τα αποτελέσματα της, της διαδικασίας του 2007. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο προτάσεις παλιότερο όσον αφορά την ισορροπία των θεσμικών οργάνων και βάση της ε, νομικής γνωμοδότησης όπου η ομοφωνία στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται σε ένα όριο του 0,03% χωρίς να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή την δυνατότητα αυτό το αυτή την προσφορά είναι κάτι που ποτέ δεν θα πρέπει να συζητήσει το Κοινοβούλιο. Το λέω ξεκάθαρα. Αναμένω το Συμβούλιο και η Κομισιόν, ιδίω όσον αφορά αυτό το άρθρο, αλλά όσον αφορά και άλλα ουσιαστικά σημεία, θα μα υποβάλει μία πρόταση για τι διαπραγματεύσει, η οποία θα συμπεριλαμβάνει αυτά τα στοιχεία και, ικανοποιητική, και θα καταλήγει σε ικανοποιητική πρόταση. Αν υπάρχει εναλλακτική για το άρθρο αυτό που μας επιτρέπει την ελόγω ευελιξία, εγώ πρόεδρε ως εισηγητής και η Επιτροπή θα ήθελα να κάνει το ίδιο, δεν θα είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω σε διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να είναι εκ των όνων κάνει. Δεν θα πάρουμε προς τα πίσω τώρα τι είχαμε πριν από 20-30 χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν αρκετές εξελίξεις θα μπορούσε να υποβληθεί μια πρόταση τον Ιούλιο με τροπολογίες και εάν δεν προχωρήσουμε θα πρέπει εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου να πούμε ξεκάθαρα απορρίπτουμε τις υποβληθήσεις προτάσεις. Θα ήταν καλό να μας καλύψει σε αυτό βέβαια η Ολομέλεια. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ο Πίτροπος Λεβατός είπε ότι η Κομισιόν δεν θα ζητήσει περισσότερες θέσεις μέχρι το 2013. Αυτό θέλω να το σχολιάσω. Δεις. Γιατί αλλού στην ημερησία διάταξη εξετάζουμε τον διορθωτικό προπολογισμό για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό το θέμα λοιπόν των θέσεων ε, απασχόλησης ε, θα πρέπει να εξετάσουμε σφαιρικά. Καλό να λέει η Κομισιόν ότι εμείς θα περιοριστούμε σε αυτά που ζητάμε και καλό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη τη σήμερα ημέρα. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε ξαφνικά να συζητάμε για κάποιες θέσεις το 2011 και δεν ξέρουμε καθόλου το 2012 και το 2013 τι μας περιμένει. Και θέλω να φέρω και εδώ αυτό που ο πρόεδρος μας ε, έχει πριστά και ε, παρουσιάσει και το έχουμε συζητήσει και με του συναδέλφου από τις Επιτροπές Προϋπολογισμών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερο τη σφαιρική εικόνα των προϋπολογισμών. Δηλαδή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης που δημιουργούμε δεν είναι η παριθμόν 28, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να συζητήσει με τα Εθνικά Κοινοβούλια να δει πού υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίες, επικαλύψεις και τι σημαίνει αυτό στο συνολική δομή του κόστους και της τοποθέτησης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τότε η δημόσια συζήτηση θα λέει ότι δημιουργούμε κάτι συμπληρωματικό στην Ευρώπη, το οποίο σε μεγάλο ποσοστό είναι περιττό. Δεν επιτρέπεται να δεχθούμε να μπούμε σε αυτή την παγίδα θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να πει ξεκάθαρα που βρίσκεται και ίσως βάσει της μελέτης που έχει παρουσιαστεί στις συνεδρίαση με τις εθνικές ε, ε, επιτροπές ε, προϋπολογισμών να εξτάσουμε λέω τι είναι σημαντικό για την εθνική δράση και τι για την ευρωπαϊκή δράση. Πέραν αυτών, εάν η Κομισιόν λέει ότι δεν θα ζητήσει κατά τα άλλα άλλες θέσεις απασχόλησης, ακόμα και αν δεν είναι δικό μου έργο, θα πρέπει να το πω. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει τότε και το Κοινοβούλιο θα πρέπει, και, και ως Κοινοβούλιο συζητήσουμε με την Κομισιόν και το Συμβούλιο κατά πόσον σήμερα επιτρέπεται μέσω ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα μπορούν να έχουν κάποια προσθέμενη αξία να υποχρεώσουμε το εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο με την εφαρμογή υιοθετημένων νόμων να πολλαπλασιάσουν τις θέσεις απασχόλησης για να εφαρμόσουν την νομοθεσία αυτή. Την σήμερα ημέρα που όλοι οι εθνικοί και περιφερειακοί προπολισμοί και όχι μόνο της Ελλάδας βρίσκονται σε μια ακραία κατάσταση από την οποία ακόμα κανένας δεν ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Και όχι μόνο οι χώρες ευρώ. Θα παραμείνουμε αξιόπιστοι μόνο εάν λύσουμε και αυτό το θέμα και αν συζητήσουμε σοβαρά πού υπάρχουν οι δυνατότητες και ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα σχέδια της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας που είναι απαραίτητα, αυτό πρέπει να αποφασίσουμε, τι θα πρέπει να αναβάλουμε και τι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τώρα. Χωρίς μια τέτοια γενική εικόνα στη συζήτηση δεν θα θεωρηθεί και το Κοινοβούλιο ως σοβαρός εταίρος. Αυτό σας το λέω εισαγωγικά. Τώρα, Ταυτόχρονα έχουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας κάποιες ώρες διατυπώσει 312, παράγραφος 3 στα αγγλικά. Το δημοσιονομικό πλαίσιο θα ορίζει όλες τις διατάξεις που χρειάζονται για την εθνική διαδικασία, ε, διαδικασία προπολογισμού για να προχωρήσει ο μελός. Και το σημείο 5 θα λέει ότι καθ' όλη τη διαδικασία αυτή το Κοινοβούλιο Κομισιών θα πάρουν όποια απαραίτητα μέτρα χρειάζονται για να διευκολυνθεί η υιοθέτησή τους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε συζήτηση αυτά που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε για τη δικασία την δημοσιονομική όσον αφορά τη δέσμη σταθερότητας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτών για μελλοντικές ε, διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό και την στάση και σχέση των θεσμικών οργάνων μεταξύ τους. Γιατί η ε, συνθήκες ισχύουν και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και για να μην ξανααντιμετωπίσουμε μια τέτοια ε, κατάσταση όπου de facto οι οι υποχρεωτικές δαπάνες, μόλις τις είχαμε καταργήσει, θα πρέπει λέω και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συνεργασία στο δημοσιονομικό τομέα στη διαθεσμική συμφωνία, θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστεί πώς θα, στο μέλλον θα αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ή και παρόμοιες καταστάσεις. Θα ήταν καλό εάν η Κομισιόν τελικά, άσχετα από το κατά πόσο νομική βάση είναι αφιλεγόμενη ή όχι, να είναι ο τίμιος μεσίτης μεταξύ των θεσμικών οργάνων και να σκεφτεί πάνω στο θέμα. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι συνεργασίες, συνεργασίες μπορούν να υπάρχουν μεταξύ αξιότιμων εταίρων εάν αυτό το θέμα δεν έχει επιληθεί επαρκώς. Και θα πρέπει καταρχήν να διευκρινίσουμε τα θέματα και θα πρέπει στην αρχή της διαπραγματεύσεων να έχουμε τις τίμιες απαντήσεις και όχι στο τέλος να τα βάλουμε όλα σε ένα τορβανά και να τα καντέψουμε. Πρόκειται βέβαια για πάρα πολλές συζητήσεις που θα έχουμε μετά την... τον ειδικό φόρου όσον αφορά τις λεπτομερείς τροπολογίες και ενδεχομένως τις προτάσεις για συμφωνίες συνεργασίας και προσαρμογή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Πρόεδρε, θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα να δούμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων ποιες είναι οι ιδέες που έχουν και ευχαριστώ να συζητήσω μαζί τους. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το εξετάσουμε αυτή τη στιγμή, να το συζητήσουμε στις 12 και 13 Ιουλίου να έχουμε μετά μια προθεσμία υποβολής τροπολογιών και μετά μάλλον στη δεύτερη ολομέλεια του Σεπτεμβρίου να πέρασε αυτό στην ολομέλεια. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά κατά πόσον οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας, βελτιωμένες ελπίζω, θα μπορέσουμε να τις θεωρήσουμε σαν βάση διαπραγματεύσεων ή κατά πόσο θα προτείνουμε στην ολομέρεια τις υποβληθήσεις προτάσεις να τις απορρίψουν καταρχήν και να ζητήσουμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο βελτιωμένες προτάσεις σαν βάση των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα έλεγα να μείνει απόλυτα ανοιχτό. Αυτή είναι η δική μου σύσταση γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσον οι εταίροι μας προτίθεται να κινηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσει εδώ η συζήτηση. Ένα μικρό σχόλιο. Ο εισηγητής μας έχει δίκιο όταν λέει ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν στις προφορικές ερωτήσεις δεν είναι οι πραγματικές. Δεν έγιναν αντικείμενο προετοιμασίας σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο μία μείζων αλλαγή που συνδέεται με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και με την οικονομική και κοινωνική χρήση που διασχίζουμε, δείχνει ότι ο συνομιλητής μας από το Συμβούλιο δεν θα είναι σε επίπεδο πρέσβεων, θα είναι η ίδια αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων. Σε επίπεδο πρέσβεων είμαστε πάντα στο μηδέν. Σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων η θέση δεν μπορεί να είναι μηδέν. Γιατί η η θέση τους θα είναι ναι αυξάνουμε τον προϋπολογισμό των κοινωνι... τον εκεί όπου υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για να λάβουμε υπόψη τις νέες αρμοδιότητες της Λισαβόνας ή πολιτική θέση μειώνουμε, πάμε στο μηδέν εκτός από τομείς στους οποίους θα πρέπει να δαπανίσουμε τα πράγματα καλύτερα. Δίδοντας ταυτόχρονα εγγυήσει ότι στα πλαίσια των πιστώσεων τις οποίες βάζουμε στον προϋπολογισμό του 11 και στους επόμενους προϋπολογισμούς μέχρι και το 13 λαμβάνουμε υπόψη μας την κοινοτική χρηματοδότηση των στόχων της Ατζέντα 2020. Σε επίπεδο λοιπόν Συμβουλίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν μπορούν να μην πάρουν θέση για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο πρέσβεων, όπως και να έχουν τα πράγματα. Μηδέν, ξεχάστε το, τίποτα κτλ. Αυτό το οποίο είναι μη ρεαλιστικό είναι ότι σε κάποιους τομείς δεν θα δαπανίσουμε περισσότερα. Προφανές είναι ότι θα δαπανίσουμε περισσότερα. Και για την Παλαιστίνη, στον τομέα της νέας εξωτερικής υπηρεσίας, για το Ιράν, για τα Βαλκάνια, για το Ιράκ, θα μας ζητήσουν περισσότερα χρήματα. Για τον ίτερ, τον, αυτόν τον αντιδραστήρα, ε, ε, λείπουν ένα με δύο δις ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Ε, για το Γαλιλαίο 100.000 ευρώ, ε, 100 εκατομμύρια συγγνώμη ευρώ σχετικά με τις αλλαγές προς το πιο πράσινο της παραγωγής ενέργειας και εκεί απαιτούνται χρήματα. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης σας θυμίζω που δημιούργησε το Συμβούλιο τον Γενάρη και για το οποίο θα πρέπει να βεθεί μια τελική νομική και δημοσιονομική λύση. Όπως και να έχουν τα πράγματα λοιπόν αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν. Οι αποφάσεις αυτές θα συνδέονται με το νέο σύστημα διακυβέρνησης της Ένωσης, το οποίο θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, βάζοντας ίσως και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στα πλαίσια του συντονισμού των εθνικών δημοσιονομικών συζητήσεων. Μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας θυμίζω, θα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο Βαν Ρομπέη στις 29 Ιουνίου για να δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνδεθεί με αυτή τη νέα πολιτική συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών στα πλαίσια της νέας πολιτικής για την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης. Λοιπόν, εκεί θα μείνουμε. Ζητώ από τους εισηγητές μόνο να μείνουν στην αίθουσα, τους συντονιστές διορθώνω και αύριο θα τα πούμε στις 9 το πρωί.